Dear colleagues, Συνάδελφοι, είναι ώρα να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. εξέταση επιστημονικών θεμάτων που, ε, για τα τρόφιμα. Αυτό θα αναπληκθεί για τις 4 Δεκεμβρίου. Μ, καθώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόθεση της χωρίς τοπολογίας δεν έχει εγκριθεί από το Κορεπέρ. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η, το σχέδιο μέσα διάταξης μπορεί να εγκριθεί με αυτή την αλλαγή και μόνον. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Πολύ εύκολο σήμερα. Πρέπει απλώς να πω ότι η διερμηνία διατίθεται σε 22 γλώσσες. Δεν έχουμε εστονικά. 21 μάλλον γλώσσες και αύριο δεν θα έχουμε ε, εστονικά και μαλτέζικα. Επίσης να προσθέσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται στο Υπάρχει, μάλλον διατίθεται στα έγγραφά της στο e-meeting και ε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Το τρίτο σημείο είναι ανακοινώσεις ε, από τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 6 Νοεμβρίου. Οι συντονιστές συστήνουν, οι συστάσεις μάλλον των συντονιστών έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και περνάμε στο σημείο 4. Μείωση των εκπομπών ρήπων από οδικά οχήματα. Όπως ξέρετε έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των ρηπογόνων εκπομπών από οδικά οχήματα. Υπάρχει πρόταση στην ε, και το κείμενο στην ημερήσια διαταξή σα, στα φακέλου σα, να δώσω το λόγο στον συγγετή, τον κύριο Άλμπερτ Ντε, για να ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το θέμα. Άλμπερτ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Τζιβάνι. Την έκθεση αυτή την ε, από τον ε, συνάδελφο του Μασούμενο, ο οποίος δυστυχώς δεν επανεκλέχθηκε και προσπάθησε να με κάνει μια εισαγωγή στο θέμα αυτό. και σε ό,τι αφορά τη μείωση των γλαμερών ε, ουσιών ε, είδα το τι προτείνεται, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές προόδους, σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών γλαμερών ε, ουσιών για τη μείωση της ρήπανσης του αέρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο, προκαλεί κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο και τις προθεσμίες για την πραγματοποίηση της μείωσης αυτής. Θα τα εξετάσουμε αυτά πιο λεπτόμερως. Στην έκθεση επίσης δεν γίνεται τοποθέτηση επαρκώς σε ό,τι αφορά τη μελέτη αντικτύπου. Και με τον πιο επικριτικό τρόπο ε, πρέπει να σας πω ότι βλέπω το θέμα των πράξεων καταξιοδότησης των εφαρμοστικών κανονισμών. Επί του περιεχομένου θα επανέλθουμε αυτά, σε αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προσθεθούν τέσσερις τομείς ε, στα πλαίσια της συναπόφασης, να πάνε μάλλον από συναπόφαση ε, στον τομέα των ε, πράξεων ε, σε ό,τι αφορά τη ύψωση τόνου, γιατί ως τώρα έχουμε στο 2,8 τόνου. και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει αυτό στην απόφαση και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές μεθανίου. Σε ό,τι αφορά το διοξιδίο του αζότου, θα προτείνω λοιπόν στην έκθεσή μου τα σημεία αυτά που σας ανέφερα να μην υπησέλθουν στον τομέα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, αλλά να παραμείνουν στην συναπόφαση από του Κοινοβουλίου. Στη συνθήκη της Λισαβόνας άλλωστε αναφέρεται ότι μόνο επουσιώδη ζητήματα μπορούν να αποφασιστούν από πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Και εγώ πιστεύω ότι στα σημεία αυτά, τα τέσσερα που σας ανέφερα, Πρόκειται για βασικές προδιαγραφές. Όλα τα υπόλοιπα σημεία με βρίσκουν σύμφωνο να μείνουν στο πλαίσιο των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα προτείνω να μπει κάτι στον εφαρμοστικό κανονισμό, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί εδώ ως κοινοβούλιο δεν συμμετέχουμε όλος διόλου. Αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται. Εδώ και 10 χρόνια εργάζομαι στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων και πάντα αυτό που προσπαθούμε είναι να παραμένει, να συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Ε, ως πολιτικοί θα πρέπει λοιπόν να εμένουμε στις πολιτικές αποφάσεις. Δεν πρόκειται να τις προασπίσουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές τις αποφάσεις. Εμείς πρέπει να το κάνουμε και γι' αυτό λοιπόν ακόμα και αν είναι τόσο τεχνική η έκθεση θα ήθελα να συνεχίσει να ασχολείται και να συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να το απαιτήσουμε. Στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση ωστόσο είναι απαραίτητο να μην υποβάλει πράξη κατά σε κάποια φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει αν συμφωνείτε ή όχι. Όταν επεξεργάζεται πράξεις κατά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ζητάμε να είμαστε εκ των προτέρων ενήμεροι για το τι γίνεται. Πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της εκάστοτε πράξης. Γιατί τότε είναι μικρότερος ο κίνδυνος και αυτό συμφέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αρνηθεί το Κοινοβούλιο να περάσει πράξη κατά εξουσιοδότηση. Ήμασταν οι πρώτοι στην Επιτροπή Γεωργίας που κάναμε αίτηση στη συνθήκη της Λισαβόνας, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, να απορριφθεί πράξη κατά εξουσιοδότηση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος ε, επανυποβλήθηκε. Χαιρόμαστε λοιπόν και επιμένουμε ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Και τώρα να ξεκινήσουμε το γύρο των σκιωδών εισηγητών. Μύρια Μτάλη από τους ευχαριστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποδεχθώ και εγώ την, Ευρωπαϊκή, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε επίσης να υποστηρίξουμε τα μέτρα που συγκεκριμένα μπορούν να περιορίσουν την εκπομπή βλαβερών ουσιών στην ατμόσφαιρα και που κατά συνέπεια θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Η ρήπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον. Και για θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και τις επιστημονικέ μελέτες, οι οποίες τι υποδεικνύουν, ότι παρά το γεγονό ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας τα τελευταία χρόνια, απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από την ολοκλήρωση της προσπάθειας σε ό,τι αφορά αυτά τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν. Υπάρχουν έντονα προβλήματα σε ό,τι αφορά την υγεία. Και αυτό κυρίως προέρχεται από τα οχήματα, τα οδικά οχήματα που εκπέμπουν πολλές ε, ουσίες επικίνδυνες μεταξύ άλλων και οξύδια αζότου, διοξίδια αζότου, αζωτούχα και το καθεξής. Κατά το παρελθόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει ορίσει τα ανώτατα όρια για τις ουσίες αυτές, για τους ρήπους αυτούς αλλά γνωρίζουμε ότι σε αστικές περιοχές υπάρχει υψηλό επίπεδο οξυδίων, του άνθρακα και αιωρούμενων σωματιδίων. Και ξέρουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Περιβάλλον, οι οδικές μεταφορές εκπροσωπούν το 42% των εκπομπών οξυδίου του αζότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρξει δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να είναι πιο αποδεκτά τα όρια των τοξικών αυτών εκπομπών, ιδιαίτερω ε, σε, ό,τι αφορά τα καινούργια οχήματα που διοχετεύονται στην αγορά, προκειμένου και να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που επιτάσσει η τεχνολογική πρόοδος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει ευελιξία σε ό,τι αφορά τα όρια βάρου και την έγκριση τύπου, προκειμένου να αποφύγουμε συστήματα διπλή πιστοποίηση για κάποια οχήματα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή και στο σημείο αυτό θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που μα είπε και ο εισηγητή Αλμπερντές, πιστεύουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή, την προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν πράξει κατά εξουσιοδότηση, γιατί πιστεύουμε ότι τα όρια βάρους μπορούν να τροποποιηθούν στον ίδιο τον κανονισμό. Συμφωνούμε επίσης σε ό,τι αφορά τα ελαφριά οχήματα και σε ό,τι αφορά τις σχετικές θερμοκρασίες. Αλλά κατά την ανάλυση του κειμένου να διευκρινίσουμε ότι δεν καταλήξαμε σε λεπτομέρειες στη μελέτη δικτύπου σε σχέση με το μέτρο αυτό. Είχαμε επίση μία πρόταση να υπάρξει ένα ξεχωριστό όριο σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντική αυτή η ρήπη. Σε ό,τι αφορά το διοξιδίου του αζότου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι τελευταίες ε, τεχνολογικές εξελίξεις και καταλαβαίνουμε ασφαλώς ότι πρέπει να διευκολύνουμε την ε, εισαγωγή στην αγορά οχημάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αόριο, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον. Έχουμε ωστόσο αμφιβολίες ό,τι αφορά τις πληροφορίες για 200 ε, ρήπους, μεταξύ άλλων και του διοξιδίου του αζότου. Θα ήθελα επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει λεπτομερώς τις πληροφορίες αυτές και να μας ε, ε, εξηγήσει ακόμα περισσότερο το κανονισμό για το διοξείδιο του άνθρακα και το, το 443 του 2009 και του 2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά, μάλλον πέρα από τα τεχνικά ζητήματα του κανονισμού μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει την ε, πρόσβαση στην ε, επιδιόρθωση και συντήρηση των οχημάτων και σε ό,τι αφορά επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν βρήκα όμως συγκεκριμένα μέτρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε επίσης η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανάλωση και τους ε, δείκτες ε, κατανάλωσης ε, καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση προτείνει τρόπους βελτίωση τη αποδοτικότητα και εξοικονόμησης 2 έω 3% στην καύση καυσίμων από παλαιά οχήματα. Ωστόσο, αυτό δεν ε, αποτυπώνεται απαραίτητα στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε και ο Άλμπερτ θα θέλαμε να εκφράσουμε ότι και εμεί συμφωνούμε ότι είναι υπερβολικό ο αριθμό των πράξεων κατά σε κάποιε περιπτώσει, όταν δεν μιλάμε για επουσιώδη στοιχεία του κανονισμού γιατί κάποια από τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με ρήπου και την εκπομπή ρήπων. Επίσης, για τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας της ατμόσφαιρας και για τη μείωση των εκπομπών ρήπων θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση το κείμενο αυτό. Να μας πει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε θα καταθέσει την επίσημη τοποθέτησή της, την επίσημη θέση της. Την περιμένουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα προκειμένου να συμμοφορθεί και η νομοθεσία προκειμένου να καταλήξουν στο τελικό κείμενο. Ευχαριστώ και τώρα για το ECR. Κύριε Ζορμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μεταρρυθμιστέ και συντηρητικοί χαιρετίζουν όλες τις ε, πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στόχο έχουν τη βελτίωση τη υπάρχουσα νομοθεσία και τη γεφύρωση των κενών και συμπλήρωση των αδυναμιών που υπάρχουν. Εντοπίστηκαν ε, κάποιες ελλείψεις της εφιστάμενης νομοθεσία ε, και χαιρόμαστε που τις επισήμανε και προσπαθεί να τις διορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά στοιχεία της πρότασης είναι πολύ θετικά. Για παράδειγμα, δεν θεωρούμε το μεθάνιο άμεσα επιζήμιο για την ανθρώπινη υγεία, παρόλο που είναι ρήπος και το μεθάνιο και αιτία ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και ο τρόπος που χειρίζεται η πρόταση αυτή το μεθάνιο στον αέρα είναι πολύ θετική. Πολύ θετικό, συγγνώμη. Επίσης, ε, συμφωνούμε με την διάθεση σε εμπορία στην ευρωπαϊκή αγορά των ε, ε, αυτοκινήτων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Και επίσης ε, συμφωνώ να έχουμε ένα, μια ενιαία έγκριση τύπου. Δεν χρειαζόμαστε δύο για την επικάλυψη των προσπαθειών. Χαιρόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητα του, του αέρα και η διαδικασία θα είναι και λιγότερο δαπανηρή για τους παραγωγού. Η ομάδα μου όμως ε, προβληματίζεται με μια σειρά προτάσεων Πρέπει να έχουμε κάποια νοτόρια για τις χαμηλές θερμοκρασίες για να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Πρέπει να εξετάσουμε πιο εξονυχιστικά τις προτάσεις. Δεν θεωρούμε ότι η τελευταία πρόταση είναι απλώς η επικαιροποίηση της προηγούμενης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να υπαχθεί η πρόταση αυτή τη κατεξοδότηση πράξη. Διαφωνούμε με τη χρήση αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα μερικέ οριακέ τιμέ που αναφέρονται εδώ, οι τιμέ στόχοι, είναι πολύ σημαντικοί. Αλλά το γεγονό ότι επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπαχθούν στι κατεξοδότηση πράξη αυτέ οι πρωτοβουλίε δεν μα βρίσκει σύμφωνο. Θα πρέπει να εξετάσουμε πιο σχολαστικά αυτό το θέμα. Γι' αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες εξηγήσει για την απομάκρυση ε, για την κατάργηση των απαιτήσεων της αμμονίας για τα βαριά οχήματα. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε το άχθος για τους παραγωγούς, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι μια καλή πρόταση και επωφελής για το περιβάλλον. Επίσης, ε, τα οχήματα φυσικού αερίου σίγουρα παράγουν και εκπέμπουν αμμονία, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα για τους φιλελεύθερους ο κύριος Τόρβατ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερα από όσα μας είπαν ήδη ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές. Νομίζουμε ότι πρέπει να δούμε τις κατεξουσοδότηση πράξεις και να προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε. Να δούμε που είναι οι μεγαλύτερες διαφωνίες ως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα για τους πρασίνους, κυρία Τέιλορ. Ο κύριος Τέιλορ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. με τις τροπολογίες ε, για, τη, για τις προδιαγραφές Euro 5 και 6 έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία για να μειώσουμε τις επικίνδυνες εκπομπές από τα οδικά οχήματα. Οι οδικές μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικής ρήπανσης που πλήττει την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Η κακή ατμοσφαιρική ποιότητα δημιουργεί περίπου, ένα, δημιουργεί περίπου μισό εκατομμύριο πρόεμους προξενεί ε, μισό εκατομμύριο πρώιμου θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία θανάτων μετά το, κάπνισμα. Ο περιορισμό λοιπόν αυτή τη ρήπανση, την πηγή τη κιόλα, πρέπει να γίνει μια προτεραιότητα για όλου. Αλλά μετά την αποτίμηση τη πρόταση αυτή τη Επιτροπή, δεν μοιάζει να δίνεται επιθυμητά αποτελέσματα Λόγου χάρη είναι καθοριστική σημασία να, να μειωθούν οι αξίες του N2, οι οριακέ αξίες στο N2. Γιατί όμως οι αξίες αυτές πρέπει να συζητηθούν, από, ε, πρέπει να συζητηθούν τους αποκλειστές πόρτες και να μην ε, συζητηθούν ανοιχτά και δημοσίως για το διοξίδιο του αζότου. Ή μέχρι το 2014 για την απόσυρση των οχημάτων έπρεπε να δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτό καθυστέρησε. Γιατί ε, αυτό που είναι ενδιαφέρον σε σχέση με την πρόταση αυτή είναι αυτά που δεν περιλαμβάνει. Και να ολοκληρωθεί η εξετασή τη. Πρέπει να δούμε την μέτρηση το, της κατανάλωσης καυσίμων και τα ισοδύναμα ε, διοξιδίου και άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Βάσει τη μελέτη αντιτύπου, τα μέτρα που καλλιεργούν την οικολογική, βιολογικότερη οδήγηση θα δώσουν κίνητρα και στι επιχειρήσει και στου ε, επιμέρου ε, χρήστε να φτάσουν σε εξοικονόμηση καυσίμων μέχρι και 2 ή 3%. Έτσι μειώνεται και το κόστος. Ωστόσο, Ο κύριος Ταγιάννη ίσως είχε θελήσει να δώσει μια ρυθμιστική ανάπαυλα στους αυτοκινητοπεραγωγούς και τα μέτρα αυτά τελικά δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή τη θητεία το Κοινοβούλιο να απαιτήσει μετρητές της κατανάλωσης καυσίμων για όλα τα επιβατικά οχήματα και τα ισοδύναμα ή, ή, να χρησιμοποιηθούν για τα υπόλοιπα οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξαιρεί τα οχήματα που καταναλώνουν φυσικό αέριο από την μέτρηση και τα μέτρα για την κατανάλωση καυσίμων. Αλλά και δεν υπάρχει σοβαρή εξοικονόμηση καυσίμων και όπως φαίνεται και από την κρίση στην Ουκρανία. Η τυπικοποιημένη χρήση φυσικού αερίου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργούμε και να το επιδιώκουμε. Η, προτιμη, η προτιμησιακή αντιμετώπιση των οχημάτων που καταναλώνουν φυσικό αέριο μειώνει και υποβαθμίζει τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ουσιαστικά παραβιάζει την αρχή της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας. Αντίκειται με τους στόχους της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο λοιπόν δεν θα πρέπει να δώσει τέτοιες δυνατότητες εξαίρεσης από τις απαιτήσει για την πρόληψη ε, και την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Επίσης, οι, το, οι συνολικές εκπομπές το THC, είναι κάτι που πρέπει να ισχύσει και για τη βενζίνη λόγω χάρη, το οποίο είναι και τοξικό προϊόν και μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η τεχνολογία για να παρακολουθήσουν τις εκπομπές THC είναι μια τεχνολογία που εδώ και χρόνια διατίθεται. Οπότε τα ε, ανώτερα όρια πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά, όχι να καταργηθούν. Τα όρια THC θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν στο δυνατόν συντομότερα. Στην ε, δοκιμή για τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυτά που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει η Επιτροπή για τα ε, οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του αζότου. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να επηρεάσει για την αλλαγή των ε, ορίων αυτών. Η αμμονία επίσης δημιουργεί προβλήματα και αναπνευστικές δυσκολίες κάτι πολύ δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα βαρέα οχήματα έχει ε, εισάγει μέσω του Euro 6 όρια για όλες τις περιπτώσεις εκπομπών αμμονίας. Αυτά τα όρια πρέπει να ισχύσουν για όλα τα είδη κινητήρων. Και τέλος για τα ελαφρά ε, εμπορικά οχήματα ή τα φορτηγάκια, αυτά που μένουν εκτός της κατηγορίας N1 και όπου δεν υπάρχει ειδική άδεια ε, ειδικό δίπλωμα οδήγηση ή ειδικά όρια με χαμηλότερα ε, ε, τέλη κυκλοφορία, εκεί βλέπουμε να υπάρχει εξαίρεση ως προς τις, τους περιορισμούς για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, τα φορτηγάκια. Μπορεί να μεταφέρουν περίπου 2,5 τόνους το πολύ. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον τα όρια αυτά να εφαρμόζονται και στην ε, πράξη. Διότι αυτή η προκατάληψη κατά των ε, οχημάτων αυτών έχει οδηγήσει σε πολύ αρνητικές συνέπειες και εμπορικές και οικονομικές και περιβαλλοντικές. Οπότε αντί να ε, μεγαλώσει αυτή η κρίζα περιοχή και να ισχύσει για τα ε, ε, ελαφρά εμπορικά οχήματα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τα πράγματα λίγο πιο σαφή. Να μην επιτρέψουμε μεγαλύτερη ευηλιξία λοιπόν για την κατηγοποίηση των βαρέων οχημάτων και των ελαφρών εμπορικών. Ευχαριστούμε τώρα για την ευθυντή κυρία Εύη. Ευχαριστώ η πρόταση που έχουμε μπροστά μας αφορά την απόφαση να ε, αναθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, αναθεώρηση κάποιων ορίων υπογόνων εκπομπών για εμπορικά και επιβατηγά οχήματα. Παρά τις αρχικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ενώ με τη γενική της κατεύθυνση συμφωνούμε, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε ότι η τελευταία νομοθετική παρέμβαση της Επιτροπής για τη μείωση των εκπομπών από τα οχήματα ε, βασίστηκε στην αντίθετη αρχή από του «οριπένων πληρώνει». Ε, επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι η ισχύουσα νομοθεσία βάσει των προτάσεων της Επιτροπής ουσιαστικά έπληξε τους μικρούς κυβισμούς ε, και τους μικρούς κινητήρες ωφελώντας τις, ε, τα μεγαλύτερα οχήματα και την κυκλοφορία τους. Η μεροληψία στις νομοθετικές επιλογές της Επιτροπής είναι κάτι που ε, δεν ε, αμφισβητείται, αλλά τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν. Τελικά τα οχήματα που δεν έχουν καλά περιβαλλοντικά αποτελέσματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Βλέπουμε επίσης οι δοκιμές των κατηγοριών 4, 5 και 6 είναι εύστοχες, αλλά χρειάζονται καλύτερη τεχνολογική διοργάνωση. Επίσης, δεν είναι σκόπιμο νομίζουμε να μεταφερθούν κατά εξουσιοδότη τη που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της πρότασή τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκλώτσα. Σας ευχαριστώ. Δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο, αλλά ο συνάδελφος Τέιλερ με προκάλεσε σε ό,τι αφορά τους ε, τα προβλήματα που έχουμε, που είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς θανάτους που προκαλούνται. Αν λοιπόν από τα μεγάλα οχήματα η συγκέντρωση σωματιδίων μπορεί να καταργηθεί, πρόκειται για ένα μεγάλο παράγοντα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση και της ρήπανση του αέρα και της υγείας. Εγώ ήμουνα το τέσσερις για το γύρο 5, γύρο 6. Και για τον λόγο που υπήρξε ειδική αντιμετώπιση ήταν οι τραγωνάνθρακες. Από... Σε μία μέρα λοιπόν καταργήθηκαν οι ρήποι αυτοί. Τα οχήματα αερίου θα είναι το ενδιάμεσο στάδιο για την ε, οχήματα δρόμων ανθρακών. Θα πρέπει και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να α, υπάρξει ανάμειξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά το e-mobility. Είναι πολύ ωραίο και καλό. Όλοι έχουμε καλή αίσθηση γιατί δεν έχουν ρήπους αυτοί, αυτά τα οχήματα. Αλλά ουσιαστικά μεταφέρουμε τους ε, ρήπους στη βιομηχανία. Υπάρχει ουσιαστικά μεταφορά των ρήπων από τους ρήπους από τα οχήματα. Θα έχουμε πιο πολλούς ρήπους βιομηχανικούς. Και πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι σημαντικό να υπάρχει η μεταβατική αυτή η φάση. Και δεν θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις τεχνολογίες αυτές. Θα είναι μια ενδιάμεση φάση αυτή σε ό,τι αφορά τα οχήματα αυτά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είτε κατά σύμπτωση είτε όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά σήμερα διαβάζουμε μία έκθεση στον τύπο του Transport and Mobility, ένα, ένας οργανισμός ε, σοβαρός από το Πανεπιστήμιο του Λούβεν για τα ηλεκτρικά οχήματα, για τα αιωρούμενα σωματίδια και τις εκπομπές τους και σε ό,τι αφορά το οξύδιο αζότου των ηλεκτρικών οχημάτων. Και ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της μελέτης, ότι η εκπομπή σωματιδίων και οξυδίου του αζότου είναι περίπου το, ίδια όπως αυτή των μικρών οχημάτων που χρησιμοποιούν βενζίνη. Τι σημαίνει λοιπόν η μελέτη αυτή, τι σημαίνει η διαπίστωση αυτή σε ό,τι αφορά και την έκθεση του κυρίου Ντές, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Αν προκύψει δηλαδή ότι η εκπομπή α, οξυδίου του αζότου είναι σχεδόν η ίδια. Και δεν μιλάμε για τις εκπομπές ε, καυσαερίων, αλλά άλλες εκπομπές που έχουν να κάνουν με τα, το φρενάρισμα, την πέδηση, με την, ε, το λιώσιμο από τα λάστιχα. Και εκεί φαίνεται λοιπόν ότι είναι ίδιες ε, οι εκπομπές και στα ηλεκτρικά οχήματα. Εγώ είμαι λοιπόν μεγάλος υπέρμαχος των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά θεωρώ ότι το, θέμα χρήζει επεξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Τώρα που Ολοκληρώνουμε, δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, οπότε να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Πέττινέλη, για να απαντήσει σε όλε τι ερωτήσει που διατυπώθηκαν από του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το σκεπτικό του κανονισμού. Ο κανονισμός περιλαμβάνει πέντε μέτρα που προσπαθούν να καλύψουν πέντε δυναμίες του τρέχοντος κανονισμού και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ατμοσφαιρικής της ποιότητας του αέρα. Τις κατατάξαμε σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε μέτρα ε, που προσπαθούν να καταργήσουν το υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθο. Το δεύτερο, δημιουργεί πιο ευνοϊκέ προποθέσει για, για οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα. Και η τρίτη κατηγορία απαρτίζεται από μέτρα που αφορούν την περιβαλλοντική απόδοση των οχημάτων. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε λοιπόν μέτρα που καλύπτουν ε, οχήματα με μεγαλύτερη μάζα αναφοράς και εκεί αποφασίσαμε να καταργήσουμε την απέτηση διπλού ελέγχου για να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία με την ενιαία έγκριση τύπου και χωρίς ε, να επιφέρουμε αλλαγές φυσικά στην ποιότητα του αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι από τις πιο σημαντικές και αφορά ε, την τροποποίηση των οριακών τιμών αμμονίας για μερικές κατηγορίες ε, οχημάτων και τη συμπερίληψη του μεθανίου στον υπολογισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αφορά μέτρα για εκπομπές οχημάτων ενώ τροποποιούμε τα, τις οριακές τιμές ρήπων για τα ελαφρά οχήματα. Και για να υιοθετήσουμε αυτούς τους στόχους και για να τους υλοποιήσουμε θέλουμε να εντάξουμε στα υπάρχοντα όρια ένα ε, όριο για τα διοξίδια του αζότου και επίσης ε, να λάβουμε υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Δεδομένων τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις που έθεσαν οι ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όντως το εγγύς μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει πρόταση μεθοδολογίας για τις πραγματικές εκπομπές από την οδήγηση και από τα οχήματα. Γιατί εκκρεμούν ακόμη κάποια τεχνικά ζητήματα, πάντως το έργο μας συνεχίζεται και θα συμπληρώσουμε τον κανονισμό για τις εκπομπές και θα το καταστήσουμε και πιο αποτελεσματικό για τις πραγματικές εκπομπές των οχημάτων θα είμαστε πολύ πιο κοντά στα όρια που προβλέπει ο κανονισμός. Υποβλήθησαν ερωτήσεις για τις πληροφορίες ε, της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. Φυσικά υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά ο βασικός όγκος αυτών των πληροφοριών θα συμπεριληφθεί σε άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τώρα υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν τους μετρητές ε, κατανάλωσης ε, των καυσίμων και κάποιους δείκτες. Δεν έχουμε περιλάβει τα δύο μέτρα στη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί η πρόταση επικεντρώνεται στα οχήματα. Άσχετα από τις συσκευές που περιλαμβάνονται μέσα. Και τη συμπεριφορά του οδηγού. Πάντως το πιο σημαντικό σημείο είναι αυτό που αφορά τα τα δικαιώματα, τι αρμοδιότητε και φυσικά το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων. Δεδομένου της ε, αναγκαίας ε, ε, ευθυγράμμιση νομοθετική που θα πρέπει να γίνει το κανονισμό 715 με τη συνθήκη της Λισαβόνα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κατάλογο με τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν κατα... καταχωρηθεί και ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ε, θέλουμε να προσαρμόσουμε τον κανονισμό 715 στις ε, νέε μα αρμοδιότητε που απορρέουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα με βάση τη διαδικασία Omnibus. Και η πρόταση καλύπτει και τα νέα μέτρα και τα υπάρχοντα που θα πρέπει να υιοθετούνται με βάση τη κατεξουσιοδότηση πράξη. Και μάλιστα η προσέγγιση αυτή συνάδει με την κοινή συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το θέμα τη έγκριση τύπου συμπεριλαμβάνεται ε, στην ε, προσέγγιση για τα διαφορετικά επίπεδα. Οπότε ένας, ένας κανονισμός συναπόφασης αφορά το πεδίο εφαρμογή οριακέ τιμές, τις ημερομηνίες εφαρμογής και εφαρμόζεται με ένα και μόνο εφαρμοστικό κανονισμό που υιοθετείται με την ε, κανονιστική ρυθμιστική διαδικασία με τον έλεγχο. Αυτή τη διαδικασία τη ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μειωθεί η γραφειοκρατία της συναπόφασης μάλλον το άχθος του νομοθέτη στα πλαίσια της συναπόφασης και να αποφευθεί η επιφόρτωση, ε, η φόρτωση μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τεχνικά ζητήματα. Αυτά και νομίζω ότι απάντησε για το θέμα των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε αυτή αμέσω στο επόμενο σημείο τη σα διάταξη, σημείο 5. αντίρρηση βάση του άρθρου 106 του κανονισμού περί οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στο, στο συνάδελφο Eckhout για να μας παρουσιάσει την ε, παρατήρηση του. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Μπάς, Θε να μιλήσει εσύ? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν το συμφωνήσαμε αυτό προηγουμένως με τον συνάδελφο, αλλά ας ξεκινήσω εγώ. Για όσους δεν γνωρίζουν για τι θέμα πρόκειται, Μιλάμε για άλλη μια επώδυνη και μακροχρόνια και κοπιαστική πρόταση με τις οποίες εργάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι νομίζει ότι μιλάμε για περιπτώσεις που αφορούν κάτι άσχετο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στον Καναδά ε, και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ πραγματικά ο στόχος είναι να υπάρξει μείωση των εκπομπών των εταιριών με χρήση διαφορετικών πηγών ε, ε, πετρελαίου, ε, παραγωγής πετρελαίου. Γι' αυτό το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ιδέα να υπάρξουν διαφορετικές τιμές για τα διαφορετικά είδη πετρελαίου, τις διαφορετικές κατηγορίες πετρελαίου. Το πιο γνωστό ήταν η πετρελοφόρος Άμος του Καναδά. Γι' αυτό μετά άρχισαν να προτίθονται και άλλα είδη παραγωγής πετρελαίου. η πρόταση του 2011 βέβαια ε, ε, σταμάτησε να εξετάζεται και μπλοκαρίστηκε στην ομάδα εργασία ε, των θεμάτων αυτών στο Συμβούλιο. Ήταν συγκεκριμένε οι χώρε, οι χώρε που είχαν πετρελαϊκέ βιομηχανίε στην εκλογική και του περιφέρειε που μπλόκαραν την πρόταση αυτή, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατοχώρε ε, με τη ΣΕΛ, η Γαλλία με την Total. Έτσι προέκυψε η αντίσταση στην πρόταση αυτή και υπήρξαν και κάποιε χώρε που απήχαν. Ε, Ένα φάκελο ο οποίο γνώρισε λοιπόν τρομερή αντίσταση παρά και την ανστήριξη που είχε από την άλλη, αλλά δεν πέτυχε την πλειοψηφία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανέπεμψε στο κοινό συμβούλιο και πέρασε καιρό μέχρι να προτείνει κάτι καινούργιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασε μια τριετία. Εάν δείτε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξαφνικά ε, λαμβάνει υπόψη διαφορετικές, ε, η κατηγοριοποίηση μάλλον των αξιών ε, έχει αλλάξει τελείω. Και αν δείτε και τα είδη όπως για την, για την πετρελοφόρο άμμο, και, τα τον υπολογισμό σε μεγατζάουλ, οι υπολογισμοί εκεί δεν έχουν αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ουσιαστικά εμέσως πια ε, στην πρότασή της ότι για τα διάφορα είδη αποθεμάτων οι τιμές είναι διαφορετικές. Αλλά όχι τα όρια. Δηλαδή, για να πετύχει κανείς το 6% περιορισμό μέχρι το 2020, έχει μια λιγότερη επιλογή στα χέρια του βάσει της πρότασης της Επιτροπής. ουσιαστικά δεν ζητά από κανένα να μετακινηθεί προς τα καύσιμα που παράγουν λιγότερο, που προξενούν διοξιδίου του άνθρακα λιγότερο, αλλά να κάνει ένα τέτοιο μίξ που να μην χρησιμοποιεί αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ε, παραγωγή εκπομπών. Είναι λοιπόν περιορισμένη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί οφείλεται και η αντίρρησή μου. Αφαιρείται μία από τις επιλογές για να επιτύχει κανείς τους στόχους το 2020. Και αυτό όντως περιορίζει τις επιλογές για τους ε, φορείς, τους παράγοντες της αγοράς. Αυτό είναι περιορισμό τη ελευθερία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι και ο λόγο που έχουμε αντίρρηση. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα εξηγήσει γιατί η επιλογή αυτή αφαιρείται εδώ και ταυτόχρονα γιατί δεν παραδέχεστε ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές ε, ε, στις εκπομπές από τα διάφορα είδη αποθεμάτων πετρελαίου. Ε, Αλλιώ, ποια είναι η αιτία που κάνετε αυτή την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, μελετώντα κανείς την πρόταση, και θα θέλα εδώ πάλι μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια ανησυχία γιατί δεν υπάρχει ούτε καν η επιλογή για τους παραγωγούς να καταγράφουν τις πραγματικές τιμές αυτή η δυνατότητα γιατί αφαιρέθηκε. Γιατί ακόμη και για τι βέλτιστε επιδόσει δεν μπορεί να υπάρξει υποβολή εκθέσεων. Να πει κανεί ότι έχει καλύτερε επιδόσει. Αυτό δημιουργεί ένα παράξενο πεδίο χωρί την επιλογή αυτή. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι δεν προβλέπεται πλέον καμία ε, παρακολούθηση και αναθεώρηση. Αυτό επίση μα παραξενεύει. Διότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και η οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης για το πακέτο το 2030 δεν αναφέρει τίποτα για τις μεταφορές. Γνωρίζουμε όμως ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων είναι ένας πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να επιδιώξει και να επιτύχει κανείς μείωση των εκπομπών των ρηπογόνων αερίων. Για τι δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πρόθεση να παρατείνει τη ζωή της οδηγίας αυτής και μετά το 2020. Τώρα δεν βλέπουμε καν τη δυνατότητα αναθεώρηση. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μάλλον σκέφτεται να μην συνεχίσει με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Γιατί καιρό θα ήταν να αρχίσετε, η Επιτροπή να μα απαντάτε και με κάποια σαφήνεια σε όλα αυτά τα θέματα. Ιδού μια σειρά από ερωτήματα που και ε, εμένα με προβληματίζουν και φαντάζομαι και άλλου συναδέλφου. Και εάν δούμε αυτή τη στιγμή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω έχει, αποδυναμώνει και Ε, μειώνει τις δυνατότητες να περιορίσει κανείς, ε, να εντείνει τις προσπάθειές του για τον περιορισμό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ακριβώ γιατί απομάκρυνε αυτές τις επιλογές. Η τελική ερώτηση επίσης είναι αν μπορείτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πείτε περισσότερα για την ερώτηση που σα επέβαλε η κυβέρνηση του Καναδά για το θέμα αυτό, για την συγκεκριμένη πρόταση. Εφόσον γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά, όπως συμπεριλαμβανόταν και το σύστημα ISDS, επίλυσης δηλαδή διαφορών του επενδυτή προς ένα κράτος, αυτό καλό θα ήταν να μας το εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί οι τιμές για την πετρελαιοφόρο άμμο έχουν ε, μειωθεί και γιατί ε, η υπόλοιπη προσπάθεια έχει αμβληθεί. Μήπως μέρος του προβλήματος είναι η συμφωνία σε βάθος και σφαιρική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Έκχο, τον συνάδελφο, για τις αγωγικές σου παρατηρήσεις. Με κάλυψε και έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε. Καταρχήν να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Η αντίρρηση δεν αφορά την ίδια την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Η αντίρρηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το άρθρο 7α από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Δεν είμαστε κατά της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Τώρα, το τελευταίο τμήμα των, του πακέτου κλίματος και ενέργειας για το 2008-2009 δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Θα πρέπει λοιπόν να, να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα, γιατί εκφράσαμε αντίρρηση κατά της εφαρμοστικής απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα μου θεωρεί ότι είναι θέμα αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής πολιτικής πρώτα απ' όλα. Και αφορά κατά βάση τη χρήση της επιστήμης και των επιστημονικών πορισμάτων ως βάση της απόφασης. Και δεν μιλάμε μόνο για τις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν το κλίμα, αλλά και τις κοινωνικές οικονομικές συνέπειες των πολιτικών μας. Τι συνέβη μετά τον Οκτώβριο του 2011 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την απόφαση της, για την εφαρμογή του άρθρου 7α της Οδηγίας για την Ποιότητα των Καυσίμων, προσέκρουσε το συμβούλιο, στο Συμβούλιο. Το βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου ήταν ότι η μελέτη επιπτώσεων δεν ήταν αρκετά διεξοδική. Τι έκανε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε νέα μελέτη επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα όμως μελέτης επιπτώσεων ε, και τα συμπεράσματα ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτή της πρώτης μελέτης λέει ότι πετρέλαιο όπως το, το σχιστολιθικό πετρέλαιο ή πετρελοφόρος άμμος έχουν πολύ ψηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις συμβατικές μορφές πετρελαίου, εξού και η ανάγκη μιας τιμή τιμής βασικής για να αποτραπεί η χρήση τέτοιων πηγών πετρελαίου στα καύσιμα. Αντί όμω να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σοβαρά τη δική τη μελέτη επιπτώσεων, λίγε εβδομάδε πριν υπέβαλε μια νέα απόφαση που αφαιρεί τελείω το θέμα αυτό από τη συγκεκριμένα στοιχεία για τις πηγές. Γιατί λοιπόν αυτή η μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια και υποτίθεται πρέπει να στηριχθείτε στη δική σας μελέτη επιπτώσεων, δεν καταλαβαίνω πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα για να υποβάλλετε την τελευταία πρόταση. Κάποιε διευκρινήσει λοιπόν θα ήθελα επ' αυτού. Τώρα έχω και μία ερώτηση προ το Συμβούλιο. Και συγχαίρω το Συμβούλιο για την παρουσία του εδώ, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε εκπροσώπηση του Συμβουλίου σε τέτοιου είδου συζητήσει. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ερώτω λοιπόν το Συμβούλιο. Τι προτίθεται να κάνει. Είδα και τη δεύτερη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το συμπέρασμα είναι ένα και το ίδιο, ότι η πρόταση του 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει αλλάξει με την τελευταία μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι θα είναι αρκετά δυσαρεστημένο το Συμβούλιο από αυτή τη μεταστροφή και φαντάζομαι θα ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στην αρχική πρόταση. Ισχύει αυτό. Επίσης, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών σχετίζεται άμεσα και με τις επενδύσεις. Πού θα επενδύσουμε τα χρήματά μας οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα που ε, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα δεν είναι έξυπνες επενδύσεις. Και αν έχουμε διαφορετική κατά βάση οριακές τιμές για σχεστολιθικό πετρέλαιο, πετρελοφόρο άμμο και άλλες μη συμβατικές μορφές πετρελαίου με υψηλή περιεκτικότητα ή με υψηλές σε διοξίδιο του άνθρακα, επιβραδύναμε ουσιαστικά τις επενδύσεις σε τέτοιες ρηπογόνες μορφές πετρελαίου. Τώρα, καταργώντας αυτήν την πρόταση, απομακρυνόμενη αυτή την πρόταση και με τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενθαρρύνουμε και πάλι πετρελαϊκές εταιρείε και άλλους επενδυτές να επενδύσουν σε πιο ρηπογόνες μορφές πετρελαίου. Ερωτώ λοιπόν και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας για την ενέργεια και για το κλίμα αν από μόνοι μας ε, θα ρίνουμε επενδύσεις στις πιο ρηπογόνες μορφές πετρελαίου, γιατί αυτό το, αυτό το αποτέλεσμα θα έχει τελευταία πρόταση. Ερώτηση λοιπόν που απευθύνεται και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις αντιρρήσεις που εξέφρασαν, στην αντίρρηση μάλλον που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πολύ ακριβείς αυτές ε, ερωτήσεις. Νομίζω ότι κάτι που θα πρέπει να πούμε αυτής εξ αρχής, γιατί αυτό το θέμα μας απασχολείται και πολύ καιρό. Όταν ξεκινάμε λοιπόν τις διαβουλεύσεις, όταν ξεκινήσαμε το 2009 τις διαβουλεύσεις, έγιναν το 2010 ε, συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη, και το 2012-2013 δεν καταφέραμε να βρούμε σε συμφωνία. Κάναμε και άλλες μελέτες και άλλες διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι έχουμε καταναλώσει πολλή ενέργεια για την πρόταση αυτή. Και πραγματικά όλοι θέλουμε να δουλειωθεί η προσπάθεια αυτή. Κατανοώ την ε, απογοήτευση, γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ σε ό,τι αφορά το πακέτο του 2008 και 2009. Αλλά τον Γενάρη που ήρθα στην Επιτροπή σας είχα υπόσχεθεί ότι η προηγούμενη επιτροπή θα υπέβαλε πρόταση. Υπέβαλε πρόταση. Και σας είπα ότι μάλλον δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η δική σας πρόταση από το προηγούμενο κοινοβούλιο. Και αυτό επαληθεύτηκε. Έχουμε λοιπόν τώρα μία στεναρή άμα, πρόταση του Συμβουλίου. Και με χαρά θα σας δώσω τις απόψεις μας για το θέμα αυτό σήμερα. Για να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτεθησαν γιατί διαγράψαμε την ε, προσέγγιση ανακαταγορία καυσίμων. Καταρχάς, όταν έγινε η μελέτη αντικτύπου, αποδείχθηκε ότι το κόστος της προσέγγισης αυτής θα ήταν ε, δυσανάλογο με τα ωφέλη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αναλογικότητα, θα πρέπει να υπάρχει αναλογική ανταπόκριση, γιατί όπως εξηγήθηκε στο πλαίσιο πολιτικής για το πακέτο του 2013, το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει να συνεχίσει στόχος μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα από τα ρηκτά καύσιμα σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά το 2020. Πέρα από το θέμα αυτό, σε ό,τι αφορά τις πραγματικές τιμές, και πάλι το εξετάσαμε αυτό πολύ στενά, το εξετάσαμε και στη μελέτη αντικτύπου, υπάρχει με μεγάλο τμήμα στις σχετικές μελέτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για τη μέτρηση των πραγματικών ρήπων. 253 400 διαφορετικά συστήματα εφαρμόζονται από τις διάφορες εταιρείε σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν προκύπτει, έχει ως αποτέλεσμα πολύ διαφορετικά στοιχεία και δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες για τα κράτη-μέλη για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες αυτές, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι υπεύθυνα για την υποβολή των στοιχείων αυτών, την συλλογή και την υποβολή των δεδομένων αυτών. Δεν ήταν αναλλαγικό λοιπόν το σύστημα αυτό και αυτό και δεν συνεχίστηκε. Σε ό,τι φορά τον Καναδά. Νομίζω ότι όλοι σε κάποια φάση τα τελευταία χρόνια μιλήσαμε με Καναδούς αξιωματούχους και σίγουρα μας παρουσίασαν πολλά επιχειρήματα, οργάνωσαν πολλά εργαστήρια, ήταν πολύ πιστικοί. Και γνωρίζουμε ότι κάποια από τα στοιχεία που έθεσαν μας βρίσκουν σύμφωνους. Συμφωνούμε ότι η πετρελαιοφόρος ε, άμμος, το σχιστικό πετρέλαιο, είναι... αλλά και το ότι το αργό πετρέλαιο έχει μια συνέχεια από τη Βόρεια Θάλασσα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι η σοβιτική Ένωση, η Νιγηρία, όπου είναι πολύ μεγαλύτερο το, το αποτύπωμα άνθρακα και τμήμα της πρότασης αυτής λοιπόν είναι ακριβώς το θέμα αυτό του αποτυπώματος σε ό,τι αφορά τον άνθρακα. Γιατί αυτό που θα ζητάμε από τα δηληστήρια του στο μέλλον είναι να υπάρχει μία βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά το εργό πετρέλαιο. Είτε είναι από τη Βόρεια Θάλασσα, είτε είναι από την Ιγυρία. Θέλουμε οι πετρελαιοπαραγωγές εταιρείε να μας δίνουν τις πληροφορίες αυτές για να ξέρουμε από πού προέρχεται το πετρέλαιο αυτό. Και ανάλογα να κρίνουμε και τις εκπομπές τους για τους ε, σκοπούς της υποβολής αναφοράς. Για το άλλο θέμα της καθοδήγησης των επενδύσεων. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Το 2009 η οδηγία για την ποιότητα των ε, καυσίμων στο, στην αιτιολογική σκέψη 9 αναφέρει στη μείωση της ε, αεροποίησης ε, καυσίμων, τη χρήση όλων των πηγών ενέργειας, τη χρήση ηλεκτρισμού, ανανεώσιμου ηλεκτρισμού και νομίζω ότι ήδη καθοδηγούμε τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή έχοντας θέσει το στόχο του 6%. Επίσης ε, όμως σας ε, είπα και προηγουμένως ότι αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι να συνεχιστεί αυτό μετά το 2020. Άρα αυτό που θα θέλαμε από το στόχο για τις ανανεώσιμες που θα τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που, ορίστηκε μάλλον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από 10 ημέρες και ε, θα θέλαμε να συνεχίσουν να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες στο μέλλον. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και για το μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Συμβούλιο έλαβε την αντίρρηση αυτή που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις 7 Οκτωβρίου τρέχοντος, Και όπω ξέρετε, βρισκόμαστε στη διαδικασία της επιτροπολογία. Αυτό που συνέβη πριν δύο χρόνια, το 2012, ήταν μπλοκάρισμα της πρότασης σε επίπεδο επιτροπή. Ε, οπότε δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Συμβουλίου ε, η πρόταση αυτή. 128 ήταν ψήφοι ψήφοι ε, υπέρ, κατά μάλλον, 128 εποχέ και 89 ψήφικα υπέρ τη προταση αυτη Οπότε η τάση προ την πρόταση ήταν μάλλον αρνητική. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια αναθεωρημένη εκδοχή τη πρόταση και στην ομάδα εργασία η πρόταση αυτή εξετάστηκε στις 8 και 21 Οκτωβρίου. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση της πρότασης τη Επιτροπής και δόθηκε δυνατότητα στις αντιπροσωπείες να ε, ζητήσουν διευκρινήσεις. Προφανώς δεν ταυτίζονται οι διάφορες θέσεις των κρατών μελών και υπήρξαν και επικριτικά σχόλια από κάποιες αντιπροσωπείς. Συνολικά πάντως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προκάλεσε άκρος αρνητικές αντιδράσεις. Θα δούμε βεβαίως. Τα σχόλια των αντιπροσωπιών επικεντρώθηκαν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος και των προθεσμιών, το θέμα της έλλειψης εναρμόνισης των διαδικασιών για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που έχουν να κάνουν με την εξόριξη πετρελαίου. Δηλαδή πώς θα καταμετράτε οι λεγόμενοι upstream emissions reductions, δηλαδή η μείωση ε, ανάντι των εκπομπών. Και επειδή υπάρχουν πολλές εταιρείες σε διαφορετικά κράτη-μέλη, μετά από την ανταλλαγή απόψεων και την αποστολή των σχολείων των κρατών μελών, η Προεδρία του Συμβουλίου ετοίμασε και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ε, ελαφρώς τροποποιημένο κείμενο. Έγιναν κάποιες λίγες αλλαγές που ξέρετε ότι στο πλαίσιο της επιτροπολογίας είναι πολύ δύσκολο να επέλθουν. Επίσης οι προθεσμίες που προισχύουν είναι πολύ περιορισμένες. Οπότε η Προεδρία απάλληψε την δυνατότητα κοινή υποβολή εκθέσεων των φορέων που εδράζονται σε διαφορετικά έχουν την έδρα του σε διαφορετικά κρατημέλη και πρόσθεσε στο κείμενο μια θεολογική σκέψη για τη δυνατότητα να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραμμές. Κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ορίζουν την προσέγγιση της καταμέτρησης, της καταμέτρησης μείωσης των upstream εκπομπών. Οι αλλαγέ, όπως είπα, είναι ελάχιστες. Το κείμενο θα υποβληθεί στην ομάδα περιβάλλοντος στις 13 Νοεμβρίου και τότε τα κράτη-μέλη θα ε, τοποθετηθούν ως προς την πρόθεσή τους στην ψηφοφορία. Για να φτάσει στο Συμβούλιο προς έγκριση το θέμα αυτό θα πρέπει όλα να έχουν ε, περατωθεί μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Πρέπει δηλαδή να έχουν γίνει όλα εντό του διμήνου που προβλέπεται για τη διαδικασία τροπολογίας. Θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί τώρα το Συμβούλιο, όμως τα σχόλια που προ στιγμή έχουμε επικεντρώνονται στο ότι το μέσο αυτό, η πρόταση αυτή, θα είχε προστιθέμενη αξία συγκριτικά με την ε, πλήρη απουσία πρότασης. Δηλαδή κάπως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να υπολογίζονται οι εκπομπές στον κύκλο ζωής ε, μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό κάνει την πρόταση αυτή σημαντική ώστε να μπορέσει τουλάχιστον σε ένα σκέλος της να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα έχουν ζητήσει το λόγο διάφοροι συνάδελφοι. Ο συνάδελφος Μπέρντερ. κυρία Μπέρντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη βαθύτερη απογοήτευσή μου και την προσωπική και των συναδέλφων για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και την φοβερή αυτή μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η πισούχος άμμος, η ασφαλτούχος άμμος είναι ιδιαίτερα ρηπογόρος. Γιατί δεν το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν το λέει καθαρά και εξάστερα. Και ακούσαμε και τα σχόλια του Συμβουλίου σχετικά. Όταν μιλούμε για τις κλιματικές αλλαγές και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε για να περιορίσουμε τις ζημίες που, στο, που επιφέρουμε στον πλανήτη, θα πρέπει να απομακρυνόμαστε κάπως από την πολιτική, παρόλο που είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να στηριζόμαστε για τέτοιες αποφάσεις στα επιστημονικά πορίσματα, που δείχνουν ότι η ασφαλτούχος άμμος, η πετρελοφόρος άμμος, είναι ο πιο ρηπογόνος τρόπος ε, εξόριξης ε, καυσίμων από το έδαφος. Και το να αγνοεί κανείς ε, την επιστήμη και να λέει ότι είναι πολύ δύσκολο είναι σαν να, ξε... να εκφυούμε τον πλανήτη ουσιαστικά. Θα πρέπει να έχουμε ψηλότερες οριακές τιμές ε, των, της, της ασφαλτούχου άμμου, από ποια πηγή και αν προέρχεται. Και όλα αυτά που λέτε ότι δύσκολο είναι να υπολογίσουμε τις κάφες και τα λοιπά, ε, ε, και πώς θα βοηθήσουμε την Ιγυρία θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να αναχαιτήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, όχι να θετήσουμε τέτοιες επονίδες στις πράξεις και να επιτρέπουμε την εξόρυξη ασφαλτούχου άμμου. Επίσης, γιατί, τι γίνεται με την Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου με τον Καναδά. Έχουμε την αίσθηση ότι η πίεση που ασκεί ο Καναδάς για την πετρελοφόρο άμμο λαμβάνεται υπόψη, παρόλο που θα έπρεπε να είναι κάτι τελείως ξεχωριστό από τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Ήταν τεράστια η πίεση του Καναδά για τη συμπερίληψη της πετρελαιοφόρου άμμου και αυτή την ευνοϊκή ρυθμίση. Φυσικά δεν θα πρέπει να κάψουμε με τα ξερά και τα χλωρά αλλά θα πρέπει να λάβουμε διαβεβαιώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα έχουμε και συμφωνία με τι ΗΠΑ στην TTIP. Δηλαδή δεν θα κάνουμε εκπτώσει στα περιβαλλοντικά, στι περιβαλλοντικέ μα προδιαγραφέ για να έχουμε πάση θυσία ε, συμφωνία ελεύθερο μπορεί. Γιατί αυτό συνέβη με τον Καναδά και με την πετρελαιοφόρο άμμο. Μπερδέψαμε την πετρελαιοφόρο άμμο στο θέμα τη ΣΕΤΑ, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τον Καναδά. Και όλα αυτά ει βάρο του πλανήτη μα. Εγώ είπα στους ψηφοφόρους μου ότι σας διαβεβαιώ ότι με τη συμφωνία TTIP δεν θα συνθηκολογήσουμε ούτε θα ξεπουλήσουμε τον πλανήτη. Αλλά πώς να το πω αυτό, με τι πρόσωπο, αν έχουμε απόδειξη περί το αντιθέτου για τη συμφωνία του Καναδά. Επίσης, το Συμφούλιο αποφάσισε για τις ε, για τους κλιματικούς στόχους το 2003 και πρότεινε μείωση κατά 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων εκπνέει το 2020. Αλλά 6 χρόνια έχουμε. Έχει νόημα να συνεχίσουμε την εφαρμογή της οδηγίας αυτής ή να πούμε ότι τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε, όπως είπε ο κύριος Κανάτη, όπως μας υποσχέθηκε ο κύριος Κανιέτο, επίτροπος, ότι από τις βασικές του προτεραιότητες θα είναι η εφαρμογή του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου για το 30. Βέβαια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να λάβουμε δεόντως υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να έρχονται πετρελοφόροι άμμο στην Ευρώπη, ασφαλτούχοι ε, και να τους αντιμετωπίζουμε σαν οποιοδήποτε άλλα βιοκαύσιμα ή πηγές καυσίμων. Επίσης, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάποια μέτρα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αν όμως εμείς πούμε όχι στην ασφαλτοχοάμμο, θα μας πούν, θα καταλάβουν ότι αυτή είναι η θέση μα. Θα πρέπει να διατρανώσουμε τη θέση μα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλα τα ποσότητα ασφαλτόχω άμμου, αλλά το γεγονό ότι επιτρέπουμε την εισαγωγή τη και δεν βάζουμε ξεκάθαρε τιμέ θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα διεθνώς. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν θέλουμε αυτό το προϊόν στην επικράτειά μας, εκτός και αν έχουμε συγκεκριμένες τιμές για το ποια είναι η επιρροή του στο πλανήτη. Θα πρέπει αυτό το μήνυμα να το στείλουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, στην, και στο Συμβούλιο. Ότι δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μπέλετ. Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν κοιμόμουν. Συνάδελφοι, δεν είναι απλό το θέμα. Κατά πρώτον, να βεβαιώσουμε από την πλευρά της ομάδας μας, και δεν είναι σαφές, ότι συμφωνούμε. Θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο μείωση των εκπομπών χάρη σε πολιτικές που αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν, αλλά θα πρέπει να επιδιώκουν ακριβώς ε, τη χρήση, την αντατική χρήση ε, συμβατικών μορφών καυσίμων και ιδιαίτερα υπογόνων μορφών καυσίμων όπως οι ασφαλτούχες ή οι πετρελοφόρες Την περασμένη εβδομάδα θυμάστε ότι είχαμε μια συζήτηση στην ομάδα για την ε, διάσκεψη των μερών και τις αποφάσεις της όπου στηρίξαμε και τη θέση του συναδέλφου Γκερμπράντη. Τώρα, εάν διατρέξουμε τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνουμε πώς αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πολιτική επιλογή που έχει γίνει είναι η απλούστερη από τις προσεγγίσεις, αλλά ταυτόχρονα οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις είναι μάλλον χειρότερες ή από σχέση με τις υπόλοιπε επιλογές που μπορούσαν να εξεταστούν και οι οποίες είχαν αποτιμηθεί και υποβληθεί στο Συμβούλιο. Οπότε η επιλογή αυτή, η συγκεκριμένη μεθοδολογία ουσιαστικά δεν κάνει διαφορά μεταξύ των διαφορών κατηγοριών καυσίμων και μεταξύ των συμβατικών ε, πηγών πετρελαίου και των ε, πετρελοφόρων άμμων. Δεν είναι τέλεια η πρόταση από την άποψη την περιβαλλοντική, προφανώς αλλά μην ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πολλές φορές ο ιδανικός κόσμος είναι εχθρός του καλού. Αυτό λοιπόν που θα χάσουμε, ε, όπως υπενήχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον απορρίψουμε την, ε, το προτινόμενο κείμενο, είναι αυτό ακριβώ. Ότι προτιμούμε να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, κάποια μεθοδολογία που μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι καλύτερο από το τίποτα για τα επόμενα χρόνια. Η μεθοδολογία λοιπόν αυτή όπως προτάθηκε ε, για επιτελεί το σκοπό της, αυτό πρέπει να διερωτηθούμε. Μπορεί να μετατραπεί σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην ευρύτερη στρατηγική μας για το 2020 και προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της ποιότητας των καυσίμων όπως έχουν οριστεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί ως τώρα και βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι νέες μέθοδοι για την υπολογισμό ε, των αερίων του θερμοκηπίου και ε, σε σχέση με τα εντατικά ρηπογόνα καύσιμα ουσιαστικά οδηγεί στην αύξηση των, ε, της παραγωγής εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και τη χρήση των πετρελοφόρων άμμων στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν θέλαμε να παραμένουμε στους στόχους της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων και την περιορισμό κατά 6% των, της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θα, υπήρχε κόστο, θα υπήρχε τέτοιο κόστος για τη συμμόρφωση που θα υποχρέωνε ε, και στη χρήση των βιοκαυσίμων και επιπλέον 4 δις ευρώ τα οποία θα πρέπει να τα επιφορτιστούν οι ίδιοι οι οδηγοί. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δικαιολογήσει αυτή την επιλογή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ροντρίγκε Ρούμπιο. Ευχαριστώ. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων στο τελευταίο τμήμα του πακέτου ενέργειας και κλίματος του 2009 ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Είναι μια σημαντική πρόταση ε, η πρόταση αυτής της γιατί μπορεί να αναχαιτήσει τις ε, εισαγωγές πετρελαίου που προέρχεται από ασφαλτόχο άμμο γιατί κατά 23% είναι πιο ρηπογόνο αυτό το πετρέλαιο από το συμβατικό. Η πρόταση του 2011 περιέχει δύο τιμές. Την προκαθορισμένη τιμή για όλα τα μη συμβατικά καύσιμα και την υποχρέωση των πετρελαϊκών εταιριών να λάβουν υπόψη τη σημασία αυτών των καυσίμων. Μετά από μια πενταετή άσκηση πιέσεων, σκανδαλώδους άσκηση πιέσεων εκ μέρου των πολυεθνικών ε, πετρελαϊκών εταιριών του Καναδά και της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την ποιότητα καυσίμων που ε, ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι των πολυεθνικών που θέλουν να, επενδύσουν στα πιο, στις πιο ρηπογόνες πρώτες ύλες όπως είναι η πετρελαιοφόρος ή άμμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έτσι μπορεί να κάνει καλύτερους υπολογισμούς ε, και να έχει ακριβή και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Αλλά ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλίωσε την πρότασή της υπό τις πιέσεις του πετρελαϊκού λόμπι. Ουσιαστικά κατήργησε την ε, υποχρέωση των πετρελαϊκών εταιριών να συμπεριλάβουν στην υποχρέωση κοινοποίηση και τις αγωγές ε, ασφαλτόχου άμμου. Οπότε δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους της οδηγίας, γιατί είναι κατά προσέγγιση ε, τα στοιχεία που δίνουν οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις ε, για, τις, ε, για τέτοια προϊόντα. Και μάλιστα έχουμε καταγγελίες από σημαντικές φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις ότι οι πολυεθνικές εταιρείες του Καναδά και των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών για να μειώσουν ε, να υποβαθμίσουν τους ε, στόχους ε, για την ποιότητα των καυσίμων. Ακόμη και η Ισπανική Πολυεθνική, η Ρεψόλ και η πιέστη οδήγησαν στη μείωση των ποιοτικών προδιαγραφών για την ποιότητα των καυσίμων. Και έτσι, χάρη στι συμφωνίε TTIP και SETA, ουσιαστικά περικόψαμε τους στόχους τη οδηγία. Μία οδηγία, αν έμπαινε κανονικά σε εφαρμογή, θα εμπόδιζε την εισαγωγή ρηπογόνου πετρελαίου από ασφαλτούχοπης είτε από τον Καναδά, είτε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, είτε από αλλού. Βέβαια, έτσι ουσιαστικά επιτρέψαμε σημαντικές επενδύσεις σε ισπανικές εταιρείες για να μπορούν να επεξεργαστούν τέτοιες μορφές πετρελαίου. Στην γενέτειρά μου, για παράδειγμα, ακριβώς μια περιοχή που είναι ήδη εξαιρετικά μολυσμένη γιατί η, ο τρόπος επεξεργασίας των, ασφα, των ασφαλτούχων άμμων είναι πολύ ρηπογόνος, πολύ χειρότερη από, από, τη, τους ρήπους που προκαλεί ε, μόλιβδος, ε, χαλκός και άλλα βαρέα μέταλλα. Επίσης, ε, η επεξεργασία κατάργωση του πετρελαίου από, τέτοιες, ε, από πετρελαιοφόρο άμμο ε, υποχρεώνει τη χρήση εξοπλισμού που ουσιαστικά αυξάνει την εθαλομίχλη και τις τοξικές ουσίες, κάτι που δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο για τον ε, πληθυσμό που διαμένει κοντά σε τέτοια δηληστήρια. Βέβαια, ε, δυστυχώς αφήσαμε ελεύθερο ξέφραγο αμπέλι στις πετρελαϊκές εταιρείες και δημιουργούμε ένα άδικο σύστημα. Και δεν απαιτούμε από τις πετρελαϊκές εταιρείες να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες για να μειώσουν τα αέρια του θερμοκηπίου. Άλλωστε και οι οδικές μεταφορές εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Και ακριβώς έχουμε ε, τις οδικές μεταφορές ως το μεγαλύτερο ε, ρηπογόνο φορέα το, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Μπαρόζο ουσιαστικά ε, δεν δέχτηκε την πρότασή μας να σταματήσει τις αγωγές ασφαλτούχου πίσας και άλλων πολύ ρηπογόνων πρώτων υλών. Λυπόμαστε για αυτή τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε δεσμευτικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των μεταφορών από το 2020. Το μόνο που μου μένει είναι να απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσουμε τους στόχους και τις υποσχέσεις που έχουμε αναλάβει και να ακούσουμε του συμπολίτε μα. Ευχαριστώ, κύριο Στόρβαλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά τη συζήτηση αυτή νομίζω ότι ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κατηγορηθεί για υπερβολική συνέπεια. Δεν μας προκαλεί έκπληξη άλλωστε. Αυτό που ακούσαμε, ότι δεν μπορούσαν να βρουν ένα κοινό παρανομαστή για το πώς θα κρυθεί η πρωτεύουσα πηγή του πετρελαίου. Θεωρώ ότι είναι μάλλον πολιτικό το θέμα αυτό. Είναι πολιτική ανικανότητα ή και διανοητική ανικανότητα. Και όχι τόσο κάτι που πραγματικά δεν μπορεί να γίνει. Εκ παραλλήλου, στο άμεσο μέλλον, ένα πλοίο το οποίο θα καταναλώνει η LNG από... θα πρέπει να αναφέρει κάθε ποντίλατο, κάθε όχημα, κάθε επιβάτη που μεταφέρει. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έντονη υποχρέωση υποβολής αναφοράς και σε άλλους τομείς όπου έχουμε πολιτικά ζητήματα λέμε «Α, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και δεν βρίσκουμε λύση». Θεωρώ ότι είναι την παλιά αυτό. Θα έπρεπε να εφεύρουμε έναν δείκτη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που επιβαρύνουν κάποια τμήματα της βιομηχανίας για να μπορούμε να προσμετράμε τις ε, εκπομπές διοξιδίου αερίου χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Να δώσω συγχαρητήρια στο λόμπι για την πετρελαφόρο άμμο. Πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι από το 2009 το πακέτο αυτό θα έπρεπε να έχει σημαντικό αντικτύπο. Πολύ πολύ αποδυναμώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο Συμβούλιο, ασφαλώς. Το αφήσαμε αυτό να χρονίσει. Εν ώψη και της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, κατά πάσα πιθανότητα. Αν όμως την απορρίψουμε, τελικά θα μείνουμε χωρίς ούτε ένα στοιχείο αν παραμείνει αυτό το στοιχείο τώρα σε ό,τι αφορά την πετρελαφόρια άμμο, θεωρώ ότι θα πρέπει να Άρα, Μεταξύ σκύλες και χάριβδες. Αυτό που είναι σημαντικό για μας ως Κοινοβούλιο, το είδαμε και στο προηγούμενο σημείο, είναι να δώσουμε όσο λιγότερα γίνεται στην επιτροπολογία. Γιατί σε τελική ανάλυση θα αντιμετωπίσουμε ένα δίλημα όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ σήμερα, όπου που κανεί δεν θέλει να ψηφίσει ούτε προ τη μία κατεύθυνση ούτε προ την άλλη. ω ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών δεν έχουμε ολοκληρώσει τι σχετικέ συζητήσει. Θα τι κάνουμε βέβαια. Αλλά όπω σα είπα συγχαρητήρια στην, ε, στο λόμπι πετρελοφόρου άμμου. Πολύ καλή δουλειά. Και είναι ντροπή και όνειρο αυτό για μα. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφο Σέικχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο διότι νομίζω ότι ήταν διεξοδική η συζήτησή μα, απλώς να επιμείνω σε ένα σημείο που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό που είπατε, αλλά το βρίσκω αρκετά προσβλητικό, για να το πω έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις απαντήσεις προς το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί Τελείω διαφορετικού τρόπου διατύπωσης για το κόστος από ό,τι στη μελέτη εντεκτύπου. Και αναπτύσσεται επιχειρήματα που λένε ότι, που, ότι προέρχονται από την μελέτη αντικτύπου. Για, τις, για τα βασικό αναλογικό κόστος και την επιλογή που είχε γίνει το 2011, την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή. Είπατε κάτι που όμω σε σχέση με τη μελέτη αντικτύπου που έχει εκπονήσει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό και αν αρχίσω να σα παραθέτω και συγκεκριμένα κομμάτια τη μελέτη αντικτύπου για να είμαστε λίγο πιο σαφεί στη συζήτηση, τι βλέπουμε. Πέραν των απαιτήσεων ε, κλπ. κλπ μέσω επιπλέον κόστος που αντικατοπτρίζει το συνολικό διοικητικό ε, κόστος για τις εθνικές αρχές, αλλά συνολικά ο φόρτος για τις εθνικές αρχές είναι αμεληταίος. Και λίγο παρακάτω, εκεί που λέμε για την τιμή καυσίμων στην ε, Αγγλία, λέγεται ότι είναι πολύ χαμηλή η αλλαγή στο κόστος που να οδηγήσει σε σοβαρές μετακινήσεις και αναδιαρθρώσεις στην αγορά. Αυτά είναι παραθέματα από τη μελέτη του αντικτύπου που μας έλεγε μόλις τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τελικά μιλά για δυσανάλογο κόστος. Μα αντιφάσκεται με τη μελέτη αντικτύπου που σας διαβάζω. Δύο τεινά λοιπόν συμβαίνουν. Ή έχετε άλλη μελέτη αντικτύπου στα χέρια σας και θα ήθελα να ξέρω πού τη βρήκατε ή ε, ηθελημένα προσπαθείτε να υπονομεύσετε τη συζήτηση για να έχετε στήριξη για την τωρινή σας επιλογή. Δεν συμβαδίζετε όμως με τη μελέτη αντικτύπου σας. Αυτό από πολιτικής σκοπιάς μπορεί να γίνεται, αλλά μην παραθέτετε τουλάχιστον τη μελέτη αντικτύπου. Είναι θέμα αρχής. Δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα κατά πρόσωπο. Και ε, η θεωρία μου για το τι συμβαίνει εδώ είναι αυτή που μόλις σας ανέπτυξα. Καλό θα ήταν να το ε, συνειδητοποιούμε όλοι μας. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Πότσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι αηδιασμένος. Πριν από δύο ή τρία χρόνια είχαμε το θέμα του γαλακτικού οξέως και τότε μειώσαμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές επειδή είχαμε υποτίθεται προβλήματα σε μια εμπορική συμφωνία με μια χώρα. Τότε ήταν τα κτηνιατρικά πρότυπα και προδιαγραφές τώρα. Αντί, ε, με τους κτηνιατρικούς ελέγχους ε, στις φαγές ε, απετράπει το θέμα αυτό, τώρα και πάλι μας ζητάτε να υποτιμήσουμε, να υποβαθμίσουμε τις προδιαγραφές μας, τις περιβαλλοντικές εν προκειμένου. Και ζητάτε να χρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη που είναι εξαιρετικά ρηπογόνος και επιζήμια για το περιβάλλον. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι απαράδεκτη και επονίδιστη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάτι θα έχει να απαντήσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και δεύτερη φορά το λόγο. Σας ευχαριστώ και για όλες τις ερωτήσει και για το feedback που λάβαμε. Νομίζω ότι καταρχάς να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε και η οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για επιτροπολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε το 2013 να λάβει, ψη... να λάβει θετική ή αρνητική ψήφο. Γι' αυτό λοιπόν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο, το οποίο και έπραξε και το Κοινοβούλιο ελέγχει την πρόταση αυτή. Ναι λοιπόν, το Συμβούλιο θα μπορούσε να καταψηφίσει την πρόταση αυτή. Αυτή ήταν η απάντηση. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξαναξεκινήσει σε επίπεδο Επιτροπής. Έχουμε πέντε χρόνια μέχρι, μέχρι ότου να χρειαστεί να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία αυτή για την ε, στόχο του 2020. Άρα θα είχαμε ακόμα χρόνο να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή αν χρειαζόταν. Νομίζω ότι κάποια, άλλα, κάποια από τα άλλα ερωτήματα έχουν να κάνουν με τον στόχο του 6% και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Τα βιοκαύσιμα σίγουρα αποτελούν μία λύση. Μία άλλη λύση θα ήταν να μειωθεί το μεθάνιο σε ό,τι αφορά την εξόριξη πετρελαίου, ο ηλεκτρισμός στα οχήματα τα δικά και ε, CNG, ε, NPG, όλα αυτά θα μείωναν το αποτύπωμα του καυσίμου αυτού. Με διάφορους λοιπόν τρόπους μπορούμε να πετύχουμε το στόχο του 6% χωρίς να εξαρτώμαστε αποκλειστικά από τα βιοκόψιμα. Είναι επίση σημαντικό να υπογραμμίσουμε το εξή. Αυτό το νομοθέτημα λύγει το 2020. Έχουμε το στόχο του 2020. Ο στόχος του 6% βασίζεται στα όρια του 2010 και αυτό που αναφέρει στον Γενάρη στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υπάρξει συνέχιση του στόχου αυτού στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό που εφαρμόζουμε είναι ένα σύστημα υποβολής αναφοράς όπου θα ξέρουμε το περιεχόμενο ανθρακά διάφορων αργών πετρελαίων που χρησιμοποιούν τα δηληστήρια. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε κατά πόσον φταίνει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Νιγηρίας, της Μορία Θάλασσας, του Καναδά και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για να δούμε κατά πόσον τα καύσιμα αυτά συνεισφέρουν ή όχι στο στόχο του 2030 για μείωση 40% σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά για το μέλλον. Και για την ανάπτυξη της μελλοντικής πολιτικής. Δεν θέλω να ξεκινήσω να μιλάω για εμπορικές συμφωνίες έτα και TTIP. Ωστόσο, ξέρω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται σχετικό πρότυπο στο, στη συμφωνία TTIP. Στην Καλιφόρνια, στη ΣΥΠΑ είναι χαμηλό το αποτύπωμα, χαμηλός ο στόχος. Και παρόλα αυτά λοιπόν υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες εφαρμογή του στόχου. Βλέπω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από πλευράς της Αμερικής σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη της διάταξης αυτή στην συμφωνία TTIP. Ο Μπάς τοποθετήθηκε πολύ στεναρά, τέλος. Και θα ήθελα να πω το εξή. Όταν μιλάω για αναλογική αντίδραση, αυτό έχει να κάνει και με το στόχο του 2020, γιατί δεν υπάρχει μετά τίποτε άλλο. Και αυτό ήταν η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το είχαμε κατά νου όταν υποβάλαμε την πρόταση. Προτείνουμε κάτι και εφαρμόζουμε κάτι το οποίο θα κρατήσει κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια. Τα κράτη-μέλη θα χρειαστούν 2 χρόνια για να το μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία. Τέσσερα χρόνια θα είναι λειτουργικό λοιπόν το σύστημα. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι αν επιβληθούν πάρα πολύ περίπλοκες διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου και διαδικασίες επαλήθευσης, δεν είναι αναλογικό αυτό σε σχέση με το τι θα επιτευχθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, υπό αυτή την έννοια μιλούσα. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη αντικτύπου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο επόμενο. Και θα ήθελα να καλέσω εδώ τους διευθυντές ε, όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών να λάβουν θέση στο Προεδρείο για να μας κάνουν τις παρουσιάσεις τους.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 Cari colleghi, così eh, Συνάδελφοι, όπως συμφώνησαν οι συντονιστές στην ε, συνεδρίαση του μηνός Σεπτεμβρίου, διοργανώνουμε μια συνεδρίαση με την παρουσία εδώ των ε, διευθυντών των οργανισμών των οποίων οι αρμοδιότητες συνδέονται στενά με τις ε, δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες της δικής μας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό διοργανώσαμε τη σημερινή συνάντηση. Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί σε μια ιδιαίτερη μορφή, διότι αποφασίσαμε πρώτα να έχουμε παρουσίαση από όλους τους διευθυντές, από τον κύριο Ντάνσα που θα παρουσιάσει γενικώ και τους πέντε οργανισμούς και μετά θα έχουμε δύο ομάδες παρουσιάσεων. Η μία θα γίνει από τον ε, διευθυντή του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και μετά από τον ε, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων. Θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις, ένας γύρος ερωταπαντήσεων και μετά μια δεύτερη ομάδα παρουσιάσεων με του διευθυντέ τη Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψη και Ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο με τον γύρο των ερωταπαντήσεων πάλι μετά. Σκοπό είναι να παρουσιαστούν οι δραστηριότητε των οργανισμών και να βεβαιωθούμε ότι όλα τα νέα μέλη τη Επιτροπή μα μπορούν να ε, λάβουν καλύτερη γνώση για τις δραστηριότητες των οργανισμών, των αρχών και των κέντρων. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε αμέσως με το Διευθυντή Ντάντσετ, ο οποίος θα μας κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους, μέλη του Κοινοβουλίου, Ήθελα εκ μέρους των ε, συναδέλφων μου και από τους υπόλοιπους οργανισμούς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω συνολικά το έργο μας. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Πρόεδρο, τον κύριο Λαβία, αλλά και τον προηγούμενο σας Πρόεδρο, τον κύριο Γκρότε, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα για αυτήν την παρουσία μας και τις παρουσιάσεις εδώ. Είμαι ο κ. Ντάντσε, ο υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και ζητήθηκα, μου ζητήθηκε και από του συναδέλφου να κάνω εγώ μια κοινή παρουσίαση. σω να είμαι ο αρχαιότερο υπάλληλο. Κάποιοι ίσω να πούν ότι είμαι και ωραιότερο και γι' αυτό αναλαμβάνω την ε, αρμοδιότητα αυτή. Θα το πείτε εσεί στο τέλο των παρουσιάσεων. Σκοπό μου είναι να σα δώσω μια συνολική εικόνα για το τι κάνουμε για τους πολίτες στην Ευρώπη να ξεκινήσω λοιπόν με μια παρουσίαση. Θα έπρεπε να μπορώ να μετακινηθώ από αυτή τη διαφάνεια. Sorry for this <laughs> technical problem. Μα συγχωρείτε για αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Ε, υπάρχουν ε, δυσκολίες με τον υπολογιστή. Επόμενη διαφάνεια ίσως. All Let me just start. Um... Να ξεκινήσω. Σύντομα θα δείτε. Α, να το. Να το βλέπετε μια πολύ, ένα πολύ απλό στιγμιότυπο. Πικνίκ. Μια οικογένεια με τους φίλους της σε ένα πάρκο. Πόσο απέχει από το έργο των πέντε οργανισμών θα σκεφτεί αυτό κανείς. Αλλά θα κάνει λάθος, γιατί αν δείτε προσεκτικά τις λεπτομέρειες της κοινής, οι άνθρωποι αυτοί τρώνε τρόφιμα που είναι ασφαλέστερα λόγω της δουλειάς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφαλεία των τροφίμων. Η κουβέρτα στην οποία κάθονται και τα παιχνίδια με τα οποία παίζει το παιδί ή τέλο πάντων τα ενδύματα που φορούν είναι ασφαλέστερα λόγω του οργανισμού για τις χημικές ουσίες που καλύπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα χημικά προϊόντα. Το περιβάλλον το οποίο απολαμβάνουν προστατεύεται από το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχετε μέτρα του στην Κοπενχάγη. Και άμα αρρωστήσουν, θα γίνουν καλά και θα πάρουν φάρμακα που θα τους θεραπεύσουν χάρη στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στο Λονδίνο. Και επίσης είναι και καλοκαίρι. Κάθονται στο γρασίδι με κοντομάνικα. Δεν βλέπετε βεβαίως τα κουνούπια που πετάνε γύρω τους και μερικές φορές και τους ε, ψήλους που, τα τσιμπούρια που είναι στο γρασίδι γύρω τους. Ο Ευρωπαϊκός, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και Έλεγχο των Νόσων στη Στοκχόλμη τους ε, προστατεύει από τα τσιμπήματα αυτά των ε, εντόμων και ο σκύλος είναι προστατευμένος χάρη στο έργο της ΕΦΣΑ στην Πάρμα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στο Λονδίνο. Υπάρχει λοιπόν προστασία για τους πολίτες, αυτούς που βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά και για εσάς και όλους τους συμπολίτες σας. Αυτό που κάνουμε πραγματικά έχει σημασία διότι διασφαλίζουμε και προωθούμε την υγεία και την ευημερία των ε, πολιτών και του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, δίνοντας ανεξάρτητες συμβουλές και πληροφορίες στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολιτικούς ηθήνοντες βάσει των καλύτερων ε, αποδεκτικών στοιχείων και επιστημονικών στοιχείων που διαθέτουμε. Το ίδιο κάνουμε και οι πέντε εδώ, ο καθένας στον τομέα του, μέσα σε διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια. Ωστόσο επιδιώκουμε κοινού στόχου. πώς προσφέρουμε ε, θετικά αποτελέσματα στους ε, συμμετέχοντες και ενδιαφερομένους ή στους ιστοτόπους βλέπουμε οι οργανισμοί μπορούν να μπλέξουν όποιον ενδιαφέρεται στο έργο τους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, διότι ακριβώς έχουμε κοινέ προδιαγραφές. Ε, φροντίζουμε να υπάρχει καλή πληροφόρηση και προσφορά επιστημονικής γνώσης σε όσους λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και να διευκολύνουμε τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τη καινοτομία ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές διεθνώς. Ε, φροντίζουμε το κόστος για τους πολίτες να είναι μειωμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει πιο γρήγορα. Πώς προσφέρουμε λοιπόν και στους ενδιαφερομένους στο δυναμικό μας, συγκεντρώνονται καλύτεροι επιστήμονες και εμπειρογνωμόνες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε τα κρατημέλη μπορούμε, μπορούν να υποφεληθούν από το υψηλότερο επίπεδο συγκεντρωμένης εμπειρογνωμοσύνης. Οι πολιτικοί θύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να, να, να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις χάρη στις ανεξάρτητες συμβουλές και πληροφορίες που προσφέρουμε. Έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση προοπτική. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε τώρα. Είμαστε ειδικοί στους τομείς μας. Μπορούμε να προσφέρουμε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των νομοθετικών πράξεων που εγκρίνεται. Εμείς δίνουμε σάρκα και οστά στις ιδέες σας. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας κατά την υλοποίηση των νομοθετικών πράξεων. Και η υλοποίηση συνήθως γίνεται από τα κράτη-μέλη και εμάς τους ίδιους σε μια κοινή προσπάθεια. Επίσης, μπορούμε να προσφέρουμε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις κατά την αποτίμηση των πολιτικών και των προγραμμάτων που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί. Οπότε έτσι υπάρχει και η αντίδραση για την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ερώτηση μπορεί να έχετε. Οπότε μην διστάζετε. Ολοκληρώνω με, αυτή, με αυτές τις φωτογραφίες των πέντε εκτελεστικών διευθυντών, οι οποίοι θα σας παρουσιάσουν τους οργανισμούς, τις, τις αρχές και τα κέντρα τους και θα βρείτε και κάποια φυλάδια έξω από την αίθουσα, από τους οργανισμούς μας, ιδίως ένα φυλάδιο με τις ε, λεπτομέρειες των στοιχείων του καθενός από τους οργανισμούς μας. Εάν πάτε στην κοινή μας σελίδα για επαφές θα βρείτε ε, τις επαφές του καθενός μας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Και τώρα να ξεκινήσουμε με, τον, με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έναν προς έναν και με τον ε, διευθυντή Hans Brunix. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, μεγάλη μου τιμή και χαρά που μπορώ να παρουσιάσω εδώ σήμερα τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Είμαστε ένα από τα πέντε ε, από τους πέντε οργανισμούς που αναφέρθηκαν. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δώσουμε σωστή και έγκυρη πληροφόρηση στους ηθήνοντες ε, και στο κοινό για θέματα περιβάλλοντος, αλλαγής κλίματος ε, και βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν λέμε στους ηθήνοντες, αυτούς που καθορίζουν την πολιτική, εννοούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, πληροφορίες, με τη Γυρωστάτα, το κοινό κέντρο, ερευνητικό κέντρο και με άλλους θεσμικούς οργανισμούς, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε 33 κράτη-μέλη, τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης και την Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Τουρκία. Προσπαθούμε λοιπόν να παρέχουμε τις απαραίτητες Στοχευμένε πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο. Πέραν αυτού, παρέχουμε διάφορες πληροφορίες και αυτό γιατί θέλουμε να σημειωθεί βελτίωση σε ό,τι αφορά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, πλαισιώνουμε την εργασία μας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τη βάση γνώσεων που υποστηρίζει αυτή τη πολιτική και θέλουμε να είμαστε η πρωτεύουσα πηγή γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών στα θέματα περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα 500 περίπου νομοθετήματα ε, του κεκτημένου του κοινοτικού κεκτημένου. Παρέχουμε λοιπόν πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, πόσο απέχουμε από τους στόχους που έχουν τεθεί, από τα πρότυπα, τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και όλο και πιο πολύ αξιολογούμε τις πολιτικές και το τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει εν ώψη και της ατζέντα και της καλύτερης εφαρμογής. Θέλουμε επίσης να είμαστε το κορυφαίο κέντρο γνώσης σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις και τους μακροπρόθεσμους στόχους και αυτό σύμφωνα με την ατζέντα για το κλίμα που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, θέλω να είμαστε η κορυφαία οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσης και, και οικοδόμησης ικανοτήτων. Και εδώ να πω ότι συνεργόμαστε με το IONET, ένα δίκτυο 39 χωρών με 1.500 εμπειρογνώμονε και με Ευρωπαίου εταίρους όπω το GRC και τη Eurostat. Επίσης συνεργαζόμαστε στενά με την υποστημονική κοινότητα με διάφορου τρόπου και το μοντέλο, το μοντέλο γνώσης και ικανότητα σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, το μοντέλο που έχουμε αναπτύξει θεωρείται υποδειγματικό. Ας εάν και άλλοι οργανισμοί έρχονται σε επαφή μαζί μας για να διδαχθούν από το δικό μας μοντέλο ανταλλαγή γνώσεων. Επίσης, να δούμε τα τρία χρονικά πλαίσια με τα οποία δομείται η εργασία μας. Καταρχάς το κεκτημένο, όπου είμαστε υπεύθυνοι για την υποβολή αναφορά σε ό,τι αφορά την ποιότητα αέρα, ε, νερού, ε, μετριασμός αντικτύπου στο περιβάλλον, μεταφορές, ε, περιβάλλον, περιβάλλον και υγεία, όλοι οι κινητήροι μοχλοί πίσω από την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτό σε ό,τι αφορά το κεκτημένο και σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορών που θα τη γνωρίζετε. Και κατά δεύτερον, επικεντρωνόμαστε στην ορία ζούντα 2020-2030 για το κλίμα και την ενέργεια, αλλά και γενικότερα για τους στόχους για το 2020 και σιγά σιγά τοπιζόμαστε προς την ατζέντα για το 2030. ποικιλία αποδοτικότητα πόρων. Θέλουμε λοιπόν να παρέχουμε γνώση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ατζέντα για το 2020-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 7ο πρόγραμμα για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος, θέτουμε και μακροπρόθεσμους στόχους σε ό,τι αφορά την ε, κυκλική οικονομία, την αποδοτικότητα και την ε, ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Προφανώς έχουμε και τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Για να δώσουμε το πλαίσιο λοιπόν, ε, ένα πλαίσιο στις προκλήσεις, χρησιμοποιούμε το εξής διάγραμμα. Έχουμε τον τίτλο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Αυτό τι σημαίνει ότι τα κοινωνιοοικονομικά συστήματα τα οποία χρειάζεται η κοινωνία μας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των πλαισίων των οικοσυστημάτων. Άρα η ποιότητα και η ποσότητα των εθνικών πόρων και των ε, στοιχείων οικοσυστημάτων είναι απόλυτα απαραίτητα ως όροι προκειμένου να δώσουμε αυτή την αξία στην κοινωνία αναδιατυπώνοντας τα κοινωνικονομικά μοντέλα και πιστεύουμε ότι αυτό είναι στο επίκεντρο της πράσινης κυκλικής ατζέντα της ε, οικονομίας και του περιβάλλοντος και είμαστε τεθειμένοι να σας υποστηρίξουμε σε ό,τι αφορά την ατζέντα αυτή. Το Μάρτιο του επόμενου έτους θα δημοσιεύσουμε επίσης μία επισκόπηση πενταετή για την κατάσταση και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, η SOER έκθεση. Βασικό δημοσίευμα αυτό, το βασικότερο δημοσίευμά μας θα αποτελείται από 87 ε, briefings 11 σελίδων για τις παγκόσμιες τάσεις, τις παγκόσμιες μεγάλες τάσεις, γιατί συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι μόνο δεν δράει η Ευρώπη σε κενό, οι παγκόσμιες τάσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και θέτουν και σύνορα και όρια σε αυτά που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, 25 θεματικές ενημερώσεις για θέματα όπως η ποιότητα του αέρα, του νερού, άλλα ενεργειακά συστήματα, μεταφορές, υγεία, αστικά συστήματα, η πράσινη οικονομία, τέτοια θέματα θα πραγματευτούμε για νέα θέματα, βιοπικιλία, γεωργία, πίεση στο περιβάλλον θα γίνει συγκριτική ανάλυση στις 39 χώρες της Ευρώπης. Και κάθε χώρα από αυτές τις 39 χώρες θα μας δώσει μία ενημέρωση αναχώρα. Επίσης για την Αρκτική, τον Εύξηνο Πόντο και το Μεσογειακό Σύστημα θα υπάρξει ενημέρωση. Τα απορίσματα από τις 87 αυτές εκθέσεις ενημέρωσης θα συντεθούν σε μία έκθεση, μεγάλη έκθεση, η οποία και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και θα γίνει, θα παρουσιαστεί αυτή η έκθεση από το Μάρτιο του 2015 στις Βρυξέλλες, μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 30 χώρες έχουν δεσμευθεί να κάνουν ε, εθνικές παρουσιάσεις των εκθέσεων αυτών. Και τελευταία διαφάνεια, να σας καλέσω όλους σας να ρίξετε τουλάχιστον μία ματιά. Αν θέλετε να γραφτείτε κιόλα στο νέο σύστημα διανομής ε, πληροφοριών. Είναι ένα σύστημα στοχευμένης πληροφόρησης, όπου κανείς μπορεί να επιλέξει τι θέλει να λαμβάνει ως πληροφορίες, για ποιους τομείς θέλει να ενημερώνεται από τους τομείς που πραγματεύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι ελπίζουμε να μπορέσουμε με τη δική σας βοήθεια να σας παρέχουμε τις ε, γνώσεις που χρειάζεται για να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις. Ευχαριστώ και τώρα θα επανέλθουμε στον κύριο Ντάνσετ. Που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. So going back to Helsinki now. Επιστροφή στο Ελσίνκι. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων είναι σχετικά νεοσύστατο οργανισμός. Δημιουργήθηκε το 2007 μετά την υιοθέτηση του κανονισμού REACH. Προηγουμένως ε, εργαζόμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ετοιμαζόμουν για την ε, ε, για τον οργανισμό αυτό. Ήταν, ήταν πολύ εντατικέ, πραγματικά οι προσπάθειε. και μάλιστα 25-35 άτομα είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον οργανισμό αυτό για να μπορεί να είναι λειτουργικό από την 1η Ιουνίου του 2007 έξι μήνε μόλι μετά την θέση σε ισχύ, την ε, έγκριση μάλλον του σχετικού κανονισμού. Τι κάνουμε λοιπόν, ε, κατευθύνουμε την εφαρμογή πραγματικά πρωτοποριακής ε, χημικής νομοθεσίας υπέρ της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας και της ανταγωνιστημότητας. Πολύ συχνά ε, ο κόσμος ε, θεωρεί ότι πρόκειται για αντιφατικούς σκοπούς, αλλά για μας δεν είναι αντιφατική, γιατί συνεχώς πρέπει να βρίσκουμε την ισορροπία να ακροβατούμε μεταξύ αυτών των στόχων κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Έχουμε και ένα πολύ γνωστό σύστημα, no data, no market, δηλαδή ε, απαγορεύονται οι μη καταχωρημένες ουσίες. Αν οι εταιρείε δεν υποβάλλουν στοιχεία και δεδομένα για τα χημικά τους προϊόντα δεν μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά, ούτε να τα κρατήσουν στην αγορά. Και λαμβάνουμε πολύ αυστηρές αποφάσεις ε, που μπορεί κανείς να τις προσβάλλει βέβαια είτε στο, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είτε στο Συμβούλιο, το εφετικό. Βλέπετε την ιστοσελίδα μας που την έχουμε οργανώσει με βάση τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Βοηθούμε τις εταιρείες να συμμορφωθούμε την κοινοτική νομοθεσία. Προσφέρουμε εργαλεία πληροφοριών και τεχνολογιών για να μπορούν οι εταιρείες να καταγράφουν όλες τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας ε, την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία και τις ε, προδιαγραφές τις καλύτερες. Επίσης παρέχουμε σωστή καθοδήγηση λεπτομεριακή στις εταιρείες για να μπορούν να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προωθούμε την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών, δηλαδή λαμβάνουμε στεναρές αποφάσεις ε, για να φροντίσουμε ότι οι πληροφορίες που, που παρέχονται είναι ποιοτικές, οι πληροφορίες είναι έγκυρες, ακριβείς και πληρούν τις προδιαγραφές της σωστής ενημέρωσης. Επίσης παρέχουμε πολλές πληροφορίες και άμεσα προς καταναλωτές για τις χημικές ουσίες και στους ε, επαγγελματίες χρήστες των χημικών. Μπορείτε να πληκτογραφήσετε το, την ονομασία οποιαδήποτε, οποιαδήποτε χημική ουσία ε, στην ιστοσελίδα και θα έχετε άμεση πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε που έχει συγκεντρώσει ο οργανισμό μα. Επίση, ασχολούμαστε και με τι ουσίε που προκαλούν ε, μεγάλη ανησυχία ή λιγότερο μεγάλη ανησυχία. Βλέπουμε ποιος είναι ο βαθμός της ανησυχίας και αν υπάρχουν περιορισμοί στις άδειε. Χρησιμοποιούμε καταρχήν αυτά τα εργαλεία σε πρώτο βαθμό, ώστε να φροντίσουμε αυτές οι επικίνδυνες ουσίες, οι ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία να χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο να αντικαθιστώνται στο, στο, στο ταχύτερο, με το ταχύτερο δυνατό ρυθμό και προωθούμε και την καινοτομία. Όπως είπα και προηγουμένως, θα διαρωτηθείτε εδώ Πού βρίσκονται τα χημικά προϊόντα, πού είναι οι χημικές ουσίες στη ζωή μας. Μα είναι μαζί μας καθημερινά και συνεχώς. Γιατί κάθε υλικό ε, αποτελείται από χημικές ουσίες. Κάθε ζωντανό όν, κάθε εμβιόν απαρτίζεται από χημικές ουσίες. Τώρα το έργο μας για τον κανονισμό REACH προσφέρει πληροφορίες, έλεγχο και ασφαλή χρήση των βιομηχανικών χημικών προϊόντων προς όφελος του περιβάλλοντος, των πολιτών και των εργαζομένων. Ο κανονισμός REACH είναι ο πιο πρωτοποριακό κανονισμό και πιο πρωτοποριακή νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα στον κόσμο. Πολύ φιλόδοξη νομοθεσία, πολύ απαιτητική για τη βιομηχανία, αλλά έχει απτά και χειροπιαστά ωφέλη και για τι εταιρείε που ενστερνίζονται το νόμο και εγκρίνουν βελτιώσεις και προχωρούν ε, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Το έργο μας για τα βιοκτώνα. Έχουμε τον σχετικό κανονισμό για τα βιοκτώνα ώστε να έχουμε έλεγχο των ε, χημικών και των κραμάτων των μειγμάτων που χρησιμοποιούν τους βιοκτώνα, όπως είναι απολυμαντικά, ε, κάποιες εντομοποθητικά ή χρώματα αντιρρυπαντικά ή άλλες κατηγορίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως βιοκτώνες ουσίες το έργο μας για τον κανονισμό CLP που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμαση και τη συσκευασία επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και η προσαρμογή του στις προδιαγραφές του ΟΗΕ. Το έργο μας ε, για το PIC, που εξασφαλίζει γνώση για, την, ε, ε, για τις εμπορικές ανταλλαγές επικίνδυνων προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και φυσικά την ευκαιρία να, που δίνουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες να πούν όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Τώρα, πού διαπρέπουμε στην εφαρμοσμένη επιστήμη, στην εφαρμογή της επιστήμης, δηλαδή διαπρέπουμε στην ε, εκτίμηση, αξιολόγηση κινδύνων και στη διαχείριση των κινδύνων όπου χρειάζεται αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης διαπρέπουμε σε έλεγχο μεγάλης κλίμακας δεδομένων και σε ανάλυση, στην εφαρμογή έξυπνων διαδικασιών με τα πιο σύγχρονα μέσα πληροφορίας και τεχνολογίας, με πληροφορίες που μπορεί να βρει κανεί επιγραμμικά και με ε, ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας, επίσης με τα, τις προδιαγραφές του ISO διαπρέπουμε και στη διαφάνεια, στο άνοιγμα που εφαρμόζουμε, στι άμεσε επαφέ με του ενδιαφερομένου και τι εταιρείε, αλλά κυρίως με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τέλος, διαπρέπουμε στην έντονη συνεργασία, εντατική συνεργασία που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, από κοινού μαζί σας προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ασφαλή χρήση των χημικών. Και βλέπετε και το σύνθημα της τελευταίας μας, μας για την ταξινόμηση των μειγμάτων μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου θα ισχύσει και θα πρέπει να γίνει αναταξινόμηση όλων των μειγμάτων από τη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2015. Και γι' αυτό έχουμε επαφέ με όλα τα κρατημέλη και μεριμνούμε ώστε όλοι όσοι υπέχουν αυτή την ευθύνη να την υλοποιήσουν και όλα. Ε, Σας ευχαριστούμε και τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Ζητώ από τους συναδέλφους που θέλουν το λόγο να τον ζητήσουν και να τον λάβουν. Ο σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση να κάνω στον κύριο Νταντσέ. Σωστά, σωστά προφέρω το όνομά σας. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν, ένα θέμα κατανόησης ε, για μια περίπτωση στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βαβαρία εμφανίστηκε. Έχουμε, έχουμε μια επιχείρηση λοιπόν η οποία ...κατασκευάζει φυσικό γυαλί και χρησιμοποιεί διάφορα χημικά, τα οποία στη τελική ανάλυση βρίσκονται στην κατάλογο των υποψήφιων ουσιών, όπως αναφέρεται. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι κατά πόσον τα χημικά αυτά θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνα, ποιες δυνατότητες υπάρχουν να συζητηθούν αυτά πιο επακριβώς, γιατί αν σωστά κατάλαβα αυτή η απόφαση δεν λαμβάνεται στο Κοινοβούλιο, αλλά πιο πολύ μεταξύ ΕΚΑ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κρατών μελών. Σας ερωτώ λοιπόν κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε άμεση επαφή μαζί σας για το πώς μπορούμε να παραπέμψουμε ενδεχομένως την σχετική εταιρεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος και τώρα έχουμε μία ερώτηση της κυρίας Σερίτ Περίκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρουσε η η παρουσίαση. Μία ερώτηση να κάνω όμως συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά την αξιόπιστη πληροφόρηση, μιλάτε για τους επιστήμονες ή και οι επιχειρήσεις, οι αγρότες για παράδειγμα. Δεν το ρωτώ αυτό τυχαία. Στην Ολλανδία αντιμετωπίσαμε περιπτώσεις όπου για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αμμονίας, αζότου κτλ. Μεγάλες επενδύσεις λοιπόν από πλευρά της Γεωργίας. Και τώρα μαθαίνουμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες δεν βοήθησαν καθόλου. Και ακούμε ότι διάφοροι κανόνες θα έρθουν από πλευρά της Ευρώπης, αλλά όλα αυτά είναι για τις θέσεις επασχόλησης. Το θέμα λοιπόν είναι θα πρέπει να είναι το περιβάλλον και έχει θέσει απασχόληση. Ρωτώ λοιπόν αληθεύουν τα στοιχεία αυτά. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο, ο κ. Ντελαφρόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια-δύο ερωτήσει για το Διευθυντή Μπρούινεκ. Ελπίζω ότι το πρόφερα σωστά. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι συγκεντρώνετε και παράγεται πληροφορίες για τους πολιτικούς και όσους ενδιαφέρονται για τα πολιτικά θέματα, για τις παραπλωτικές ε, πολιτικές και τα παραπλωτικά θέματα. Και κάτι μας είπατε και για την ε, αποστολή και την ε, κυκλοφορία των πληροφοριών που αποστολούνται σε πολλές χώρες και τη συγκεντρώνεται και από πολλέ χώρε. Μπορείτε να μα πείτε ποια είναι συγκεκριμένα τα εργαλεία με τα οποία μεταδίδεται όλε αυτέ τι πληροφορίε σε εμά σε εμάς που εργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα. Ε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο πέραν των ενδιαφέρουσων δημοσίευσεων που κάνατε. Τι άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται και επίσης υπάρχει και η αντίστροφη ροή. Δηλαδή μπορεί κανείς να αποταθεί στον οργανισμό σας όταν εργάζεται επί συγκεκριμένων θεμάτων ή φακέλων για να έχει συγκεκριμένες απαντήσεις για κάποιο θέμα. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριο Τάι. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους ε, τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Δύο ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Ταρσέτ. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δεδομένων και των φακέλων ε, καταχώρησης, αυτό μας απασχόλησε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το 2012, τον Μάιο του 2012, ο κύριος Τεχρότε ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος μετά από, τους τονιστές, από αίτημα των συντονιστών σας απέστειλε μια επιστολή για την ποιότητα. Κάντε λοιπόν ανακοινωθέν τύπου τον Ιανουάριο του 2014 μετά από αξιολόγηση του 5% των φακέλων που είχαν να κάνουν με την προθεσμία του 2010 για διάφορες ουσίες, μεγάλο όγκο χημικών, χημικά, πάνω από πάρα που είναι πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, για καρκινογόνες, ουσίες, ε, ουσίες που προκαλούν ε, μεταλλάξεις και διαπιστώνουμε, διαπιστώνεται ότι στο 79% των φακέλων δεν υπάρχει συμμόρφωση, ότι υπάρχουν δηλαδή ε, ελλείψεις. για μεγάλο ποσοστό των ουσιών μιλάμε. Και αυτό προκαλεί ανησυχίες και για το περιβάλλον και για τα τρόφιμα, την ασφάλεια τροφίμων. Θα συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι η συμμόρφωση των θεμάτων αυτών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δράσης αυτής και της, ε, του οργανισμού σας που πραγματικά λειτουργεί καλά, αλλά πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά. Πώς θα φροντίσετε λοιπόν τα θέματα αυτά, τα εφάκελοι καταχώρησης να είναι επαρκής, γιατί αν 69% δεν στέκει, θεωρώ ότι είναι προβληματικό το ποσοστό αυτό. Κατά δεύτερον, η όλη συζήτηση Πελάτες. Πολύ επικίνδυνο για την αναπαραγωγική υγεία. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση με την βιομηχανία που λέει ότι υπάρχουν υποκατάστατα της ουσίας αυτής, κυρίως ε, στο PVC χρησιμοποιείται, αλλά υπάρχουν διάφορα προβλήματα υψηλής τοξικότητας και ερωτά η βιομηχανία. Κατά πόσον είναι προβληματικό το ζήτημα αυτό. Κάποιες φορές λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν ως επιχείρημα την τιμή, το κόστος που είναι πάρα πολύ ψηλή, διατείνεται η βιομηχανία. Εσείς λέτε ότι ο οργανισμός σας θα δώσει έγκριση στο προϊόν αυτό, βάσει των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Θα ήθελα να ξέρω, τα επιχειρήματα αυτά στέκουν ή είναι δικαιολογίες προκειμένου να χορηγηθεί τελικά η επιστοποίηση ή έγκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Γκρότε. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς χαίρομαι που τα καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την ε, συνεδρίαση, γιατί θεωρώ ότι οι οργανισμοί έχουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για την αιμοθετική μας εργασία. Έχουμε συναντηθεί τακτικά και τα άτομα επαφή. Ε, που συμμετείχαν στην αποστολή και που δώσαν αναφορά εδώ στην Επιτροπή μας ε, ήταν πολύ χρήσιμα και έχουμε και νέους συναδέλφους εδώ μαζί μας σήμερα οι οποίοι ενδεχομένως να κατανοήσουν έτσι τη μεγάλη ποικιλία των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για θέματα περιβάλλοντας αντίθετα με τα εθνικά κοινοβούλια για το γερμανικό κοινοβούλιο μπορώ να σας πω όπου έχουμε επιστημονικές υπηρεσίες οι οποίες ε, είναι σε φάση κατασκευής. Αυτό που μας ε, δίνουν όμως οι οργανισμοί αυτοί για το νομοθετικό μας έργο είναι ανεκτήμητης αξίας και σήμερα βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου πραγματικά. Και εδώ γίνονται και ακροάσεις, ε, όπως τους επίτροπες, όταν ορίζουμε τους εκκληστικούς διευθυντές, κάνουμε συζητήσεις και το Κοινοβούλιο παρακολουθεί το τι κάνουν οι οργανισμοί. Ωστόσο, οι οργανισμοί αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Γι' αυτό έχει σημασία να το τονίζουμε και να το υπογραμμίζουμε. Γιατί στη δημόσια συζήτηση πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό, το παραμελούμε. Να καλέσω λοιπόν τους συναδέλφους, τους νέους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν τους οργανισμούς. Σίγουρα υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχει και κριτική σε πολλές περιπτώσεις όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά πάρα πολλά επιτέχθησαν τα τελευταία χρόνια. Όταν μιλάμε για το ρίτς και το κατηγορούμε, για παράδειγμα, αλλά από την άλλη όταν πρόκειται για θέματα χορήγησης προϋπολογισμού σφίγγουμε τα ζωνάρια και κάνουμε περικοπές. Δίνουμε πιο πολλές αρμοδιότητες δηλαδή στους ορισμούς, αλλά δεν τους δίνουμε χρήματα. Αυτό είναι αντιφατικό αυτής εξ αρχής και τότε να μην παραπονιόμαστε στην τελική ανάλυση. Αν θέλουμε να κάνουμε περικοπέ εδώ πέρα, να έχουμε υπόψη είναι ότι αν υπήρχαν 28 διαφορετικέ τέτοιε υπηρεσίε, τα πράγματα αυτά είναι πολύ πιο ακριβά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν του οργανισμού αυτού στη τελική ανάλυση. Και όχι να κάνουμε περικοπές όταν καθορίζεται ο προϋπολογισμός και μάλιστα περικοπές που δεν έχουν κανένα νόημα. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για λεφτά φορολογουμένων αλλά θα πρέπει να έχει νόημα η εργασία τους και θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να εξοικονομούμε χρήματα. Γι' αυτό χαίρομαι λοιπόν που έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Giovanni Λαβία την ευκαιρία αυτή σήμερα να εξοικονομουμε χρηματα γι αυτο χαιρομαι λοιπον που εδωσε ο προεδρος της επιτροπης γιωβανη λαβια την ευκαιρια αυτη σημερα να κανουμε μια συζήτηση με τους ε, επικεφαλής των οργανισμών. Και θα μπορέσουμε φυσικά να συνομιλήσουμε και κατηδίαν με τους επικεφαλείς. Ευχαριστούμε. Ματίας ο κύριος Φλόρενς. Αυτό που είπε ο κύριος Γκρότε, το υπογραμμίζω και εγώ επισταμένος. Πολύ λυπάμαι που τα αποτελέσματα των οργανισμών σπάνια, πολύ σπάνια τελικά επηρεάζουν το πολιτικό έργο. Και στην περίπτωση αυτή δεν απαλλάσσω για τον εαυτό μου, θα ήθελα να ενισχύσουμε τους οργανισμούς θα πρέπει να φροντίσουμε τα αποτελέσματα όμως, τα πορίσματα, να καταλήγουν και μέσα στα κεφάλια των συναδέλφων. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει αποτελέσματα, να μην είναι χωρίς ε, χρήση τα πορίσματα αυτά. Κάτι άλλο τώρα. One Substance, One Registration. Πριν από την ψηφοφορία χιλιάδες σελίδες ήταν το έγγραφο αυτό και ήταν ε, η άγκυρα σωτηρίας για τα κρατημέλη. Τώρα λοιπόν ε, πάτωσε αυτή, μάλλον η πρόταση αυτή δεν έσωσε κανέναν. Γιατί τόσο άσχημα τα πήγε, γιατί πήγε τόσο άσχημα αυτή η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να υπάρχει μία έγκριση ανά και δεύτερη ερώτηση, αρκετά απλή. Από τους υπεύθυνου ε, ανακύκλωσης ακούμε πάντα ότι μετά την ανακύκλωση απορριμμάτων η πρώτη ύλη πάντα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία REACH. Στέκει αυτό. Αν έχει περάσει κάποιος τη διαδικασία REACH για μια τηλεόραση όταν θα υπάρξει ανακύκλωση τη τηλεόραση, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ήδη περάσει το ανακυκλωμένο προϊόν τη διαδικασία REACH. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον αντιπρόεδρο ο κύριο Ποτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είναι μεγάλη μα χαρά να σα έχουμε εδώ. Και χρειαζόμαστε όλο ένα περισσότερε συζητήσει και διάλογο με του οργανισμού. Διότι ήδη από την πρώτη διαφάνεια φωτογραφία που μα δείξατε Όλα δείχνουν ειδηλιακά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και όλοι είμαστε συνεχώς ασφαλείς και προστατευμένοι. Όμως δεν αληθεύει αυτό, γιατί τους μεθόδους, τις μεθόδους για την δοκιμή των ε, μακροχρόνιων χημικών ουσιών τις περιμένουμε, όπως και επίσης για τη μακρά έκθεση σε ε, χημικές ουσίες, για τις αναμίξεις και ούτω καθεξής. Πάντως, όταν ήμουν εισηγητής για τα θέματα των επεκτατικών ειδών, Ήλπιζα να έχω κάποιο συνομιλητή και από του οργανισμού εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε τέτοιο διάλογο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη σαφήνεια για τι αρμοδιότητε των οργανισμών σα. Και μερικέ φορέ έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Κάποιες φορές έχει χρειαστεί να περιμένουμε πενταετία ή εξαετία για την ε, καλή προσφορά ειδικών γνώσεων ε, σε συγκεκριμένα θέματα που τα λάβαμε μετά από πέντε χρόνια για ε, συγκεκριμένες οδηγίες για, τους, για τις ενδοκρινικές ουσίες λόγου χάρη. Το ίδιο. Δεν είναι λοιπόν όλα τόσο χαροπά. Βεβαίως σέβομαι την επιστημονική σας γνώση που βασίζεται σε γεγονότα και αποδεκτικά στοιχεία. Αλλά δεν μπορούμε εδώ να αρχίσουμε να βγάζουμε γιασμό ενώ μυρίζει θείο. Ε, είναι και μια βασική αρχή των χημικών ενώσεων αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ναι, για σκοπούς ε, οικονομίας χρόνου θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η πρώτη ερώτηση αφορά το πώς ε, διαμορφώνεται η λογοδοσία μας και αν είναι αληθινά τα όσα λέμε αν βασιζόμαστε μόνο σε επιστημονική γνώση. Να πω όχι, δεν βασιζόμαστε μόνο σε επιστημονικές γνώσεις. Η δουλειά μας βασίζεται σε πολλές διαφορετικέ πηγές. Μία από τις βασικότερες είναι ότι όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις, τα monitoring στην Ευρώπη, την ποιότητα των υδάτων λόγω χάρη και το καθεξής, τα συγκεντρώνουμε και ε, μεταφέρονται στις βάσεις δεδομένων μας με μαθηματική ακρίβεια. Για, τις ποιότητα, τον έλεγχο ποιότητας δημιουργούμε δείκτες, χρησιμοποιούμε πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα και συνεργαζόμαστε με το κοινό κέντρο ερευνών και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δύο βασικά σετ επιστημονικών κριτηρίων που χρησιμοποιούμε. Έπειτα, ε, βρισκόμαστε στην εμπροστοφυλακή της καινοτομίας, ιδίω ιδίως όταν μιλάμε για αυτό που έχει ονομαστεί επιστήμη των πολιτών. Λόγω χάρη, μία εφαρμογή για τα κινητά που να συνάδει και με την πολιτική για τις ε, θάλασσες και πολίτες να βλέπουν λόγω χάρη τι θερμοκρασία επικρατεί και τι καιρό στις διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες. Αυτό είναι προσφορά πληροφορίας πολύ διαφορετική από, το κλασικό, από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε με το κλασικό επιστημονικό νου. Επίσης για τις πληροφορίες προς τις εταιρείε προσφέρουμε τέτοιες ε, πληροφορίες, αξιοποιούμε δεδομένα από τις επιχειρήσεις και τις εταιρείε. Η απάντηση είναι ναι σε περιορισμένο βαθμό. Ε, ο έλεγχος ποιότητας ε, γίνεται πάλι με βάσει τα ίδια κριτήρια και πρότυπα που εφαρμόζουμε. Εάν συγκεντρώσετε, αν δείτε τη συνολική εικόνα από όλες αυτές τις διαφορετικές πηγές, ε, έτσι ε, εφαρμόζουμε το πρόσωπο, το πρότυπο που σας είπα και αξιοποιούμε πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται για τις μελέτες αντικτύπου. Δηλαδή βλέπουμε τι πληροφορίες λάβαμε, ε, αξιολογούμε την κρισιμότητά τους και τα συνδέουμε με συγκεκριμένα θέματα. Δεν περιεριζόμαστε μόνο σε επιστημονικά απορίσματα τα οποία δημοσιεύονται σε επιστημονικά δημοσιεύματα. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα ε, πηγών επιστημονικής γνώσης. Ένα από τα στοιχεία που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός διαφάνειας σε οποιαδήποτε έκθεσή μας. Εάν ε, κάνετε κλικ σε ένα link ε, μπορείτε να δείτε κατευθείαν την πηγή από την οποία προέκυψε η μελέτη. Οπότε κρίνετε εσείς οι ίδιοι ε, εάν τα συμπεράσματα ή η αξιολόγησή μας είναι ορθά. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος βαθμός διαφάνειας. Η δεύτερη ερώτηση ήταν το πώς επικοινωνούμε ε, και πώς μεταδίδουμε τα συμπεράσματά μας. 40 εκθέσεις τον χρόνο δημοσιεύονται. Ε, δημοσιεύονται στον τύπο υπάρχουν εβδομαδιαίως. Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, όλο ένα για περισσότερο, ε, με πολλούς followers με αυτούς που μας παρακολουθούν. Επίσης έχουμε κοινέ παρουσιάσεις του έργου μας, πολλές φορές εδώ στις Βρυξέλλες. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και του Κοινοβουλίου. Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Και ε, οι συνδρομές που προσφέρουμε αυτό το ανέφερα στην τελευταία μου διαφάνεια. Αυτό σα επιτρέπει να παρακολουθείτε συστηματικά το έργο μας. Επίσης έχουμε ένα αυξημένο αριθμό έναν αυξημένο όγκο πληροφοριών επιγραμμικά online στο διαδίκτυο. Δηλαδή, όποιο θέλει να βρει πληροφορίε στο διαδίκτυο, αυτομάτως θα τις λαμβάνει και μάλιστα επικαιροποιημένε. Μπορούν έτσι και οι πολίτες και οι πολιτικοί ηθήνοντες να δουν με απόλυτη διαφάνεια το τι κάνουμε. Για την ερώτηση εάν θα μπορούσαμε να σας απαντήσουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, να πω χωρίς να κατονομάσω κάποιον, ότι σήμερα κάποιος που ήδη έχει λάβει το λόγο εδώ, πριν από δύο εβδομάδες, πριν από μια δημόσια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, ήρθε σε επαφή με τον οργανισμό μας για μια σειρά από ερωτήσεις που τον απασχολούσαν συγκεκριμένα και εντός 24 ώρου έλαβε ένα πακέτο απαντήσεων προς του ε, που έφτασε στο γραφείο του. Οπότε προφανώς έχουμε τη δυνατότητα αυτή και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας φυσικά να στηρίξουμε το έργο των βουλευτών. Οπότε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε. Τελευταία ερώτηση για τα επεκτατικά, για, για τα χωροκατακτητικά ε, είδη. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη εκδοχή της ε, πρότασης και ξέρετε ότι το άλλο σκέλος της πρότασης ε, ε, πήγε, σε άλλο εταίρον μας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και από τον οποίο περιμένουμε τις μελέτες οικοτόπου και του συστήματος. Πάντως ναι, είμαστε στην πρώτη γραμμή συλλογής πληροφοριών. Σε ευχαριστώ. Και τώρα λόγω στον κύριο Τάντσετ για να απαντήσει στις ερωτήσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση από τον Βαβαρό συνάδελφο τέθηκε. Δεν την κατάλαβα. Χειροποίητο το γυαλί. Ναι, όντω, εδώ μπορεί να έχουμε πολλές χημικές ουσίες. Ε, για παράδειγμα, τα χρώματα, οι βαφές που χρησιμοποιούνται για το γυαλί. Η μόλιβδος που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο γυαλί είναι όντως ε, ουσίες που μπορεί να συνδέονται με την πρόκληση ασθενειών. Και στο παρελθόν εργαζόμενοι στον τομέα αυτό παραγωγή γυαλιού αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας. Και μια εταιρεία που χειρίζεται ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για να δει τι μπορεί να κάνει και μάλιστα και πριν τη λήξη των προθεσμιών. Να υποβληθεί σε περιορισμούς ή ε, να ζητήσει αδειοδότηση. Αυτό είναι ένας τρόπος να έρθει απευθεία σε επαφή μαζί μας για να ενημερωθεί η εταιρεία. Τέτοιου είδους πάντως εταιρείε συνήθως ε, μπορούν να λάβουν πληροφορίες και από άλλες ε, εταιρείε του ίδιου κλάδου που ήδη διεκπαιρέωσαν με επιτυχία τη διαδικασία, δηλαδή αντικατέστησαν χημικές ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία με άλλες ουσίες που δεν είναι προβληματικές. Δεύτερη ερώτηση για την ποιότητα των δεδομένων. Ιδιαίτερα στην πρώτη προθεσμία της καταχώρησης που είναι τα χημικά με το μεγάλο όγκο. Ε, με πολύ προσοχή και σύνεση επιλέγουμε τους φακέλους για την εξέταση της ποιότητας και εκεί διαπιστώνουμε ε, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και για αυτές λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις. Και όταν λέω με ευφύ και συνετό τρόπο επιλέγουμε τα ντοσιέ, σημαίνει ότι διαλέγουμε τα ντοσιέ που ξέρουμε ότι παρουσιάζουν ε, αδυναμίες συμμόρφωσης, γιατί επικεντρωνόμαστε στις χειρότερες περιπτώσεις, εκεί που υπάρχει παραβίαση και φυσικά λαμβάνουμε αποφάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν και παρακολουθούμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι αποφάσεις μας. Και έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους του κλάδου ότι θα ξεπεράσουμε και το 5% στα χημικά μεγάλου όγκου. Συνεχίζουμε τις έρευνες για την ποιότητα αυτών των καταχωρήσεων προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές. Στο DDHIP, τους θαλάτες δηλαδή. Και αυτοί, οι θαλάτε υπόκεινται στην ανάγκη αδειοδότησης. Όσες εταιρείες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ουσίες πρέπει να λάβουν άδεια προηγούμενη. Να υποβάλουν δηλαδή αίτηση άδεια και φυσικά θα πρέπει να εγκριθεί η αίτηση αυτή και να δοθεί η άδεια. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, λίγες, γιατί οι περισσότερες εταιρείες ήδη έχουν αντικαταστήσει τις ουσίες αυτές από άλλες λιγότερο επικίνδυνες. Για παράδειγμα είχαμε μία περίπτωση άδεια που πέρασε από τις επιτροπές μας και έχει αποσταλεί με επιστημονικές συμβουλές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε τελικό βαθμό αρμόδια για τη λήψη της απόφασης. Και εδώ πάντως θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί αν δοθούν αυτές οι άδειες θα έχουν χρονικό ορίζοντα, χρονικό περιορισμό και η προθεσμία που δίνεται στις περιπτώσεις αυτές είναι μικρότερη από τις άλλες περιπτώσεις ίδιας ουσίας γιατί λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν θεωρούμε ότι τέτοιου ίδιου άδεια θα πρέπει να ισχύει για μακρά περίοδο. Βέβαια, οι επιστημονικές επιτροπές προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και υποβάλλουν τα πορίσματά τους, τα οποία σεβόμαστε φυσικά και παραπέμπουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επιστημονική Συμβουλή. Σε ό,τι αφορά τις διαρωτήσεις του κυρίου Φλόρεντς, γιατί δεν βοηθά τις μικροπαιστές επιχειρήσεις, το όζορ. Το όζορ δεν ήταν εφεύρεστα κάτι που προέκυψε στην πορεία της διαδικασίας και φαίνεται ότι δεν αξιοποιούν το όζορο τόσο όσο θα περιμέναμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τώρα που φτάνουμε στην τελευταία προθεσμία, τελικά εξαφανιστεί από την αγορά αυτό το σύστημα όζορ, μία καταχώρηση, μία για κάθε ουσία. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα περιμένουμε την αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση. Προς το παρόν δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα παραπάνω. Για την ανακύκλωση, δεν χρειάζεται πάντα η νέα καταχώρηση. Έχουμε δώσει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές και συμβουλές προς τις εταιρείες πότε χρειάζεται να κάνουν καταχώρηση μετά την ανακύκλωση. Και αν χρειαστεί καταχώρηση γιατί πρόκειται για μια ε, σχετικά νέα ουσία, τότε αυτές οι εταιρείε συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τη βασική ουσία που έχουν ανακυκλώσει. Συνήθως πάντως η διαδικασία ανακύκλωσης δεν παρενοχλείται ή δεν επιβαρύνεται ή δεν επιβραδύνεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη ομάδα οργανισμών. Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και να δώσω το λόγο στον κύριο Ούρλ, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καλησπέρα. Κυρίε και κύριοι, και από δική μου πλευρά σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σα παρουσιάσω και την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα ουσιαστικά μόνο. Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και το τρίτο και πιο βασικό, τι αξία μπορούμε να έχουμε, να προσθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων. Για το πρώτο ερώτημα. Θα ήθελα να το θέσω ως εξή. Η ΕΦΣΑ είναι ένα κέντρο ικανοτήτων σε ένα δίκτυο κρατών μελών, εμπειρογνωμόνων και μεταξύ των, Ευρωπα... των κρατικών κέντρων αξιολόγησης κινδύνου. Πολύ σημαντικό πόρισμα. Αυτό είμαστε τμήμα ενός δικτύου. Η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την υποστήριξη των κρατών μελών. Και αυτό λοιπόν καταχωρήθηκε στον κανονισμό ίδρυσης της ΕΦΣΑ, όπου και αποφασίστηκε η λήψη αποφάσεων, η συλλογή δεδομένων, η εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου θα πρέπει να γίνεται κεντρικά από ένα οργανισμό στην Πάρμα. Αλλά οι εμπειρογνώμονες παραμένουν σε επίπεδο κρατών μελών στα πανεπιστήμια, στους οργανισμούς έρευνα, στους οργανισμούς αξιολόγησης κινδύνους και η ΕΦΣΑ χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρογνωμοσύνη μέσα ανοιχτών ετοιμάτων και έτσι συνενώνεται όλη η γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα οργανισμό σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου για την διατροφική αλυσίδα η δεύτερη, το δεύτερο πρόσωπο της ΕΦΣΑ. Είμαστε πάροχος ανεξάρτητων και ε, τεκμηριωμένων επιστημονικών στοιχείων. Παρέχουμε δηλαδή στους πολιτικούς και στους ζητήνοντες τεκμηριωμένες πληροφορίες για να λαμβάνουν τις αποφάσεις της. Κάτι άλλο ότι που μάθαμε είναι ότι η αξιολόγηση κινδύνου και η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να γίνονται από άλλα να διαχωρίζονται. Άρα δεν εγκρίνει η ΕΦΣΑ τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, δεν δίνουμε εγκρίσεις γενικότερα. Το τρίτο σκέλος, το τρίτο πρόσωπο της ΕΦΣΑ, είμαστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση για τους κινδύνους. Τα θέτουμε όλα αυτά σε ένα πλαίσιο. Τα πληροφορούμε τους πολιτικούς, τους εμπλεκόμενους φορείς, διεξαγάγουμε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με το ευρύτερο κοινό, το οποίο είναι και δύσκολο, γιατί μιλάμε για 500 εκατομμύρια καταναλωτές και σε διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, με διαφορετικές γλώσσες, άρα δεν είμαστε σε θέση να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με 500 εκατομμύρια καταναλωτές και πάλι χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη Τι κάνουμε λοιπόν. Η ΕΦΣΑ κάνει αξιολόγηση κινδύνου πιστοποιημένων προϊόντων πριν την έγκρισή του. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε υπόψη μας για παράδειγμα τα πρόστιμα, τα, ένζυμα, τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζημα, τα χρωστικές, ε, αρωματικά, όλα χρειάζονται πιστοποίηση. Πριν προσθεθούν στα τρόφιμα όμως χρειάζεται και αξιολόγηση ασφάλειας. Η αξιολόγηση ασφάλειας αυτή γίνεται από τους επιστήμονες της ΕΦΣΑ, από επιστήμονες τους οποίους έχουμε βάλει στα πάνελ μας και καλύπτουμε ε, την ευημερία των ζώων, την ασφάλεια των ζώων, την ασφάλεια των φυτών, βιολογικούς κινδύνους, πρόσθετα τροφίμων, καλύπτουμε όλη την διατροφική αλυσίδα. Και αυτό ήταν συνέπεια της διατροφικής κρίσης της δεκαετίας του 90 και εφαρμόστηκε ε, αυτό ως αρχή στην ίδρυση της ΕΦΣΑ. Επίσης αξιολογούμε το κατά πόσον υπάρχει θέμα υγείας για διάφορα προϊόντα. Ξέρουμε όλοι ότι διάφορα στοιχεία των τροφίμων κάνουν καλό και ότι αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται με επιστημονικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν το κάνει η ΕΦΣΑ. Πέρα από τα πιστοποιημένα προϊόντα κάνουμε γενική αξιολόγηση κινδύνου τονίζοντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη σαλμονέλα. Η ΕΦΣΑ έχει κάνει πολλή δουλειά από κοινού με τα κράτη-μέλη, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της σαλμονέλα. Και αυτή η κοινή προσπάθεια στέφτηκε με επιτυχία, γιατί τα κρούσματα σαλμονέλας περιορίστηκαν κατά 50% και άνω τα τελευταία πέντε χρόνια. Άρα οι κοινέ προσπάθειες κατά μελών Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΦΣΑ πραγματικά είναι πολύ αποτελεσματικές. Πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε βέβαια, αλλά σίγουρα υπήρχαν αποτελέσματα στις προσπάθειές μας. Ύστερα, το κάτι άλλο το οποίο είναι στο DNA αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι στη ΣΕΦΣΑ η δημιουργία ενός δικτύου για την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Δεν μπορούμε με τα άτομα που απασχολούμε στην Πάρμα να τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Χρειάζεται ένα δίκτυο με του εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Και εδώ θα ήθελα να, το, να υπογραμμίσω το εξή. Υποστηρίζουμε όσου είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εθνικό επίπεδο. Σε διαχείριση κρίσεως και σε περίοδο διαχείρισης κρίσεων η ΕΦΣΑ μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κρίσεων αυτών. Τώρα, η προστιθέμενη αξία του οργανισμού μας. Νομίζω ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και τα πιο δύσκολα στοιχεία είναι ότι, ότι μπορούμε να συνενώσουμε όλο το εύρος των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, τους καλύτερους, να δημιουργήσουμε μια βάση γνώσης για όλα τα κρατημέλη και για τα πιο μικρά κρατημέλη που δεν θα μπορούσαν από μόνα τους να συλλέξουν όλη αυτή την εμπειρογνωμοσύνη. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι έκανε πραγματικά ένα βήμα μπροστά μπροστά. Γιατί αυτή η εμπειρογνωμοσύνη δεν διατίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Είμαστε ένα κεντρικό σώμα για τους κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων. Δηλαδή, εξοικονομούμε πολλά χρήματα στους φορολογούμενους, γιατί κάποιες διαδικα... όλες αυτές τις διαδικασίες γίνονται μία φορά και όχι 28. Και έτσι έχουμε το ίδιο επίπεδο υψηλής προστασίας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θεωρώ ότι ο νομοθέτης το 2002 όταν ιδρύθηκε η ΕΦΣΑ το έβαλε στον κανονισμό τον τρετικό και έτσι ήταν ένα τεράστιο βήμα αυτό για να εγγυόμαστε το ίδιο επίπεδο υψηλής ποιότητας προστασίας για όλους τους πολίτες. Αυτές λοιπόν οι γνώσεις ε, φυσικά διατίθενται και στους πολιτικούς, στην ε, Πολιτική Επιτροπή της ΕΝΒΗ στο Κοινοβούλιο και είμαστε ασφαλώς στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε με την παρουσίαση ε, του κυρίου Σπρίγκερ για, τον Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να βρούμε τη σωστή φωτογραφία. Γιατί με αυτή την ωραία φωτογραφία ξεκινήσαμε, αυτή την ωραία εικόνα. Αλλά εγώ θα σας μεταφέρω σε μια άλλη εικόνα. Βλέπετε εδώ μια παραγκούπολη της Μονράβια, της πρωτεύουσα της Λιβυρίας. Πολλές οικογένειες συνοστίζονται στην στη φτωχογειτονιά αυτή, σε πολύ μικρές καλύβες, δεν έχουν καν τρεχούμενο νερό και αυτή είναι η πρώτη γραμμή της καταπολέμησης του ιού έμπολα. Και πολλές από τις αναφιόμενες απειλές προέρχονται έξωθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλό θα ήταν να το συνειδητοποιήσουμε. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα της επιδημίας έμπολα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ πιο λεπτομεριακά σε αυτό το θέμα της έμπολα γιατί δείχνει ε, και περιγράφει το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου. Στόχος μας είναι να παρακολουθήσουμε, να εκτιμήσουμε και να δώσουμε στοιχεία για επιλές στην ανθρώπινη υγεία και για λοιμώδη νοσήματα. Και επίσης ελέγχουμε και ερευνούμε ε, νοσήματα γνώστου προέλευσης. Παρέχουμε ε, κατευθυντήριε γραμμές και τεχνική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και στηρίζουμε τα κράτη-μέλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τεχνογνωσία και κατάρτιση και επιμόρφωση για να προετοιμαστούν σε εθνικό επίπεδο κατά εμφάνισης ε, ακρουσμάτων ή επιδημιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιό έμπολα. Στα αρχικά στάδια οι εμπειρογνώμονές μας απλώς παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις πληροφορίες για το έμπολα που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν όταν είχαμε κάποια μηδρά ε, στοιχεία από τη Γουινέα. Κάναμε τότε μια αξιολόγηση και στις 22 Μαρτίου επιβεβαιώθηκε ότι ε, η νόσος αυτή είναι όντως ε, η νόσος από τον ιό του έμπολα. Είχαμε 90 περιπτώσεις και 60 θανάτους. Και μέσα σε 24 ώρες ε, συντάξαμε μία ε, ραγδαία ταχεία εκτίμηση κινδύνου. Και για την περίπτωση κρουσμάτων που θα μεταφέρονταν από τη Γουινέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα πολύ γρήγορα αναβαθμίσαμε την αξιολόγηση αυτή του κινδύνου και δώσαμε αυτές τις πληροφορίες και συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους είχαμε ήδη εμφάνιση του έμπολα σε πολλές χώρες. Είχαμε κρούσματα στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβυρία και τη Γουινέα. Και μάλιστα εκδώσαμε και νέα μελέτη κινδύνου, εκτίμηση κινδύνου και μάλιστα άμεσης, άμεση ε, επίπτωση. Και μάλιστα κάναμε και μια σύντομη απογραφή των ικανοτήτων των κρατών μελών να κάνουν διάγνωση του έμπολα, γιατί δεν είναι εύκολη η διάγνωση του ιού έμπολα. Οι εμπειρογνώμονές μας, μάλιστα, κατέγραψαν πληροφορίες για Ευρωπαίους ε, πολίτες που ταξιδεύουν από και προς τις χώρες που παρουσίασαν αιστείες του ιού αυτού και έτσι με τις πληροφορίες αυτές ε, καταλήξαμε στο διασυνοριακό σοβαρό χαρακτήρα που είχαμε και μάλιστα μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου αναθεωρήσαμε την ε, μελέτη κινδύνου πέντε φορές και μάλιστα είχαμε και περιπτώσεις υγειονομικής εκένωσης υπηκών Ευρωπαίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, θεραπεία. Και μάλιστα είχαμε και μια, ένα κρούσμα μιας νοσηλεύτριας που προσβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ φρόντιζε έναν ασθενή που έπασχε από έμπολα. Και μάλιστα έχουμε και δύο σε διασκέψεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Υγείας και Ασφάλειας για την Υγεία με θέμα το έμπολα και συμμετείχαμε και εμείς. Επίσης ε, έχουμε ένα δίκτυο 40 εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με το έμπολα. Κάθε εβδομάδα προσφέρουμε συμβουλές και τεχνική αρρωγή που μας ζητά τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης αποστέλουμε εμπειρογνώμονές μας σε μεμονωμένα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσουμε. Και επίσης αποστέλουμε εμπειρογνώμονες και σε διεθνείς αποστολές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για παράδειγμα. Και μάλιστα έχουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης για τα κρούσματα έμπολα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και έχουμε και τεχνικά έγγραφα και κατευθυντήρες γραμμές για μεθόδους υγειονομικής εκένωσης με ασφάλεια και επίσης για ε, το θέμα της, ε, ε, του ελέγχου εσόδου και, εισόδου και εξόδου και επίσης έχουμε και ένα εγχειρίδιο με συγκεκριμένε πρακτικές συμβουλές. Βλέπετε εδώ, δεν είναι καθόλου εύκολο να φορέσει κανείς και να ή να αφαιρέσει τον εξοπλισμό. Γι' αυτό και έχουμε δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το φόρεμα και την αφαίρεση αυτής της στολής, αυτού του εξοπλισμού. Όλες αυτές τις πληροφορίες ε, τις ε, κάνουμε και τις δίνουμε σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχουμε ξεκινήσει και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, ώστε να μπορούμε να αποσπάσουμε προσωπικό και να το μεταθέσουμε προκειμένου να ασχοληθεί με την κρίση του έμπολα. Και είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι πέρα του έμπολα παρακολουθούμε και 50 άλλες ε, νόσους, που είναι σημαντικές, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις. Ε, ε, μικροβιακή αντοχή, ε, ιός, θυματίωση, ασθένειες που αντιμετωπίζονται με εμβολιασμό και το καθεξής. Είμαστε Έχουμε συνεργασία τώρα με τα κράτη-μέλη. Έχουμε δύο μέλη μας που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τρεις από τρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καθηγήτρια Μαλιόρη και ο Καθηγητή Χίρε είναι ε, τα διορισμένα μας μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε και έναν πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελική μας έκθεση από τη δεύτερη ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση. Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη αυτή η έκθεση, αλλά πριν από λίγε εβδομάδε, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ε, αντίγραφο αυτής της ανεξάρτητης εξωτερικής ε, αξιολόγησης. Εκεί αναγνωρίζεται το κέντρο μας ως πρωτοποριακή οργάνωση για την παροχή επιστημονικής συμβουλής και καλής ποιότητας πληροφοριών, που είναι αρκούντος ανεξάρτητο κέντρο. Επίσης, το επιστημονικό του κύρος ε, ακολούθησε την ανιούσα, αυξάνεται σταθερά τον τελευταίο καιρό και μάλιστα έχει εδρεωθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα ε, μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας παντού στην Ευρώπη. Και μάλιστα το κέντρο μας είναι ιδιαίτερα υπερήφανο για τα εγκόμια αυτά της ανεξάρτητης εξωτερικής έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην τελευταία παρουσίαση του τελευταίου οργανισμού, «Έμα» και μετά και να δώσω το λόγο στον κύριο Ράζιν. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και καμάρι που μπορώ ως τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό ελπίζω, να σας παρουσιάσω τον οργανισμό μας, τον οργανισμό για τα φάρμακα. Ξέρω ότι πολλοί μας γνωρίζετε καλά, όμως για κάποιους ίσως είναι ενδιαφέρον να μάθετε κάποια στοιχεία παραπάνω για μας. Καμιά φορά όταν ε, σε κανέναν καφέ με ρωτάνε τι ακριβώς κάνει ο αίμα. Ε, θα ήθελα να πω σε μια πρόταση ότι είναι ο οργανισμός που αξιολογεί τα νέα φάρμακα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαιώνεται ότι θα είναι αποτελεσματικά καλής ποιότητας και ασφαλή προτού αρχίσουν να τα συνταγογραφούν οι γιατροί προς τους πολίτες παρακολουθεί όλα τα φάρμακα, όχι μόνο τα καινούργια, για, από την σκοπιά της ασφάλειας και ε, γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τους 28 εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων. Με μια πρόταση αυτό θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην ερώτηση τι ακριβώς κάνει ο αίμα. Όμως, πώς το επιτυγχάνουμε. Το σύνθημά μας, επιστήμη, ιατρική υγεία, ε, είναι αναφέρει τρεις πυλώνες που έχουν να κάνουν με την συλλογή επιστημονικών στοιχείων για τα εγκεκριμένα φάρμακα. τα οποία πρέπει να ε, είναι τα καλύτερα δυνατά ε, που θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Πώς θα πετυχαίνουμε αυτό. Το στοιχείο της επιστήμης στη διαδικασία του έργου μας. Συγκεντρώνουμε την καλύτερη επιστημονική γνώση ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους εθνικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, παντού στην Ευρώπη και έχουμε ε, ένα δίκτυο 3.500 ε, εμπειρογνωμόνων και ειδικών που συνεργάζονται παρασότερο στην ε, πραγματικότητα ανεξάρτητων επιστημόνων άνευ συμφερόντων οι οποίοι Διορθώνονται σε 7 ειδικέ ε, επιτροπέ, κάθε μια στο πεδίο αρμοδιοτήτων του και ειδικευσή του και σε κάθε επιτροπή το κάθε καντοσμένο έχει τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο. Δι' αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ειδικές, ειδική καθοδήγηση και επιστημονικές συμβουλές στους ερευνητές και μπορούμε να στηρίξουμε την καινοτομία, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις οποίες συμβουλεύουμε και επειδή έχουν λιγότερε ρυθμιστικέ δυνατότητε οι ίδιε. Βάσει αυτών των ε, επιστημονικών στοιχείων ε, προχωρούμε και σε συστάσεις για την έγκριση ή την απόσυρση κάποιων φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα νέα φάρμακα ή τουλάχιστον τα νέα φάρμακα για συγκεκριμένες νόσους αξιολογούνται σε κεντρικό επίπεδο, στο Λονδίνο, για νέες αγωγές όπως για το AIDS, τον καρκίνο, το διαβήτη, τις κλίσεις καταπλάκας και το Alzheimer's. Ειδικότερα μας απασχολούν τα φάρμακα που απευθύνονται σε παιδιά και οι σπάνιες νόσοι. Εργαζόμαστε βάσει μιας απλής αρχής. Μία αίτηση, μία αξιολόγηση, μία αδειοδότηση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν με το ίδιο όνομα και τις ίδιες πληροφορίες για τους γιατρούς, τα φαρμακεία, τις νοσοκόμες θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ανά την Ευρώπη. Δηλαδή ισχύει ένα πρότυπο για όλους τους Ευρωπαίους ασθενείς. Δουλειά μας είναι να εξισορροπήσουμε το όφελος και τον κίνδυνο, όχι μόνο τη στιγμή της αδειοδότησης και έγκρισης, αλλά αυτός ο λόγος πρέπει να αξιολογείται διαρκώς και στην πραγματική ζωή μετά την έγκριση ενός φαρμακού προς την ποιότητα, την ασφάλεια και προκειμένου να γίνει αυτό Όλα αυτά γίνονται βάσει της προσέγγισης δικτύου, η φαρμακοεπίβλεψη, η όπως λέγεται. Μια από τις βασικές μας αρμοδιότητες. Τώρα με την, με την υγεία τι ακριβώς γίνεται. Ε, προσπαθούμε να έχουμε καινοτόμα φάρμακα και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν ε, ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται. Ιδίως για τις σπάνιες νόσους και τα παιδιά που δεν έχουν ε, τις βέλτιστες δυνατότητες στα χέρια τους. Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε όλες οι διαθέσιμες επιλογές να διατίθενται και για τα ε, κατοικίδια ζώα, τους εκτροφείς ζώων, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε με πολύ ταχείς διαδικασίες που να καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις υπάρξει παραμικρή ανησυχία για την ασφάλεια, την ποιότητα ενός φαρμάκου, αν υπάρξει το οποιοδήποτε περιστατικό οπουδήποτε στην Ευρώπη, σημαίνει ότι είμαστε σε θέση αυτό να το μεταφράσουμε σε μέτρα ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Οπότε, νομίζουμε η δουλειά μας επιτρέπει ε, να καταλήξουμε σε αυτό το στιγμιότυπο που είδατε στη φωτογραφία στην αρχή. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνοι μας φυσικά. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς και τις ε, αδερφούς οργανισμούς Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Πρέπει να ε, ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό μας χρειάζεται περισσότερο και η συνεισφορά των ασθενών. Πρέπει να αυξήσουμε τις επιλογές αγωγής και θεραπείας που προσφέρονται για συγκεκριμένε νόσους. Γι' αυτό χρειάζεται και η καινοτομία. Ξέρουμε ότι η βιωσιμότητα και οι τιμές ε, αρχίζουν να γίνονται φραγμός για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Γι' αυτό δημιουργούμε γέφυρες για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις τεχνολογίας υγείας, για να δούμε δηλαδή το λόγο ε, ωφέλους ε, κινδύνου ως φαρμάκου αλλά το 65% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη δεν παράγονται στην Ευρώπη. Οι ρυθμοί και ε, τάσεις παραγωγής αλλάζουν. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε και τη διάσταση τη διεθνού συνεργασίας. Το είδο των ειδικών γνώσεων που χρειαζόμαστε. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την ανατεχνολογία, τη γενετική μηχανική και άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι διαρκώς πρέπει να επικαιροποιούμε τις ειδικέ γνώσεις, την ομάδα των ειδικών μας. Και ούτως ή υπάρχουν όλο ένα εντυνόμενες απαιτήσει. Πρέπει λοιπόν αυτή η διάσταση της παρακολούθησης της ασφάλειας να ενισχυθεί. Και βεβαίως θέλουμε να μας εμπιστεύονται σε αυτά που κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει τα δεδομένα μας να μεταδίδονται όσο και να διαδίδονται στο δυνατόν περισσότερο, ε, καθώ και οι σχετικές μας αποφάσεις. Γι' αυτό αυτό θέλουμε να υπάρχει και μεγάλος βαθμός διαφάνειας. Όλα αυτά σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Εδώ έχουμε πολύ καλά παραδείγματα επιτυχημένης ε, συνεργασίας με τους συναδέλφους και να θα πρέπει εδώ να αναφέρω και την ε, συμβολή των συναδέλφων στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε να πάμε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα σας ζητήσω να είστε πολύ σύντομοι, διότι έχουμε οκτώ ε, παρεμβάσεις και έχουμε και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε με την κυρία Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους διευθυντές των οργανισμών Θεωρώ ότι το έργο των ε, οργανισμών είναι κέριο, πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη λειτουργία των διαφόρων κλάδων, ιδιαίτερα για την έρευνα. Όλοι οι οργανισμοί έχουν στενές σχέσεις και δεσμούς με τους επιστημονικούς κύκλους. Εγώ γνωρίζω κυρίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, αλλά φαντάζομαι και άλλοι οργανισμοί ίδια προβλήματα έχουν. πρόσφατα ακούμε για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, όχι τόσο για τους επιστήμονες, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Και αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ίσως χρειαζόμαστε σαφέστερους κανόνες γιατί συνήθως προσάπτουμε τη σύγκρουση φερόντων σε κάποιον που έρχεται από τη βιομηχανία, αλλά όχι από κάποιον που είναι μέλος μη κυβερνητική οργάνωσης, γιατί ένα μέλος οργάνωσης κατά των γενετικών στροπημένων λογαριασμών δεν θεωρούμε ότι έχει σύγκρουση φερόντων, ενώ κάποιος που έχει δουλέψει σε συναφή βιομηχανία αμέσως του κολλάμε τη ρετσινιά τη σύγκρουση συμφερόντων. Το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων είναι κάτι που υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Αλλά θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Κάποιο που μόλι αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά κάποιο που εργάστηκε σε ένα διαφορετικό κλάδο εμπίπτει στον ορισμό τη σύγκρουση συμφερόντων. Είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο το θέμα και πιστεύω ότι χρειάζεται μια καλύτερη νομοθετική οριοθέτηση. Ένα άλλο θέμα που αφορά και πάλι την Ευρωπα... τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια των Τροφίμων. Η σχέση με του ετούντε. Ιδιαίτερα στο θέμα των ισχυρισμών για την υγεία. Οι ετούντες παραπονιούνται για την έλλειψη διαλόγου και διαβούλευσης με τον οργανισμό ΕΦΣΑ και παραπονούνται γιατί δεν υπάρχουν απλοί κανόνες για τους ισχυρισμού. Και δεν είναι εύκολο να, κάνει, να προσθέσει κανείς χειρισμούς Θα πρέπει αυτό το θέμα να το διευκρινίσουμε για το θέμα κυρίως των ισχυρισμών υγείας. Επίσης για τα έξοδα των οργανισμών. Ο οργανισμός των ε, φαρμάκων λαμβάνει κάποιους ε, δασμούς. Ε, είδαμε και το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης, αλλά δεν έχουν αυτό το προνόμιο όλοι οι οργανισμοί, πως θα πρέπει να το γενικεύσουμε για όλες τους οργανισμούς. Η κυρία Μελχιόρ, αλλά πραγματικά θα, θα σας θέρμα παρακαλούσα να είστε λακωνικοί για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Να προσπαθήσω, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους οργανισμούς που μας παρουσίασαν το έργο του σήμερα γιατί για μένα ως ε, νέο μέλος και για όλους τους νέους συναδέλφους είναι μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσουμε όλους μαζί. Σας ευχαριστώ. Δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γκούλ. Στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Είπατε ότι επί της αρχής υποστηρίζετε και τις επιστημονικές ε, τις επιστημονικές γνώσεις και ότι συνεργάζεστε με τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητα του στην ΕΦΣΑ και παράλληλα μοιράζονται τα απορίσματά τους με τα κράτη-μέλη και ύστερα τι γίνεται αν δεν υπάρχει ευρία επιστημονική βάση για την ανατοχνολογία για παράδειγμα, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και κατά δεύτερον, Δεύτερη ερωτήση. Οι πληροφορίες σας ε, πώς διατίβονται στο ευρύ κοινό. Είναι σημαντικό αυτό για την κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Όσλιν. Ο κύριος Όσλιν, σας ευχαριστώ και εγώ να ρωτήσω την ΕΦΣΑ. Ξέρετε ότι συχνά υπάρχει κριτική ότι η επιστήμη είναι πολύ κοντά με τη βιομηχανία. Έχετε προβλήματα τέτοια ανεξαρτησία. Και αν ναι, πώ θέλετε να τα αλλάξετε αυτά. Ο συνάδελφο Γκρότε είπε ότι πολλά έχουν αλλάξει και αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το θέμα που επικρίνεται. Ε, δεύτερο θέμα, μακροπρόθεσμες συνέπειες των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Πάντα υπάρχει κριτική για τη μεθοδολογία διεξαγωγής αναλύση κινδύνου. Θα αλλάξετε κάτι λοιπόν στο θέμα αυτό για τη διαδικασία επιστοποίησης που θα αλλάξει κιόλας. Τρίτη ερώτηση. Μπορείτε να αξιολογήσετε το θέμα της σχετικής μελέτης για την ουσία 810. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πιέγα. Σας ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις για τον οργανισμό, προς τον οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που αντιμετωπίζει πολύ άριθμες προκλήσεις, όπως μας περιέγραψε και ο Πρόεδρος. Ε, εμένα με ενδιαφέρει η συνεργασία με τις 27 εθνικές υπηρεσίες και την ΕΜΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, γιατί τι χαρακτήρα έχει ε, ο Οργανισμός Φαρμάκων έχει ρόλο επιτήρηση ή συνεργασία. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερη συνεργασία. Έχει βέβαια και νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Τα βιοτεχνολογικά φάρμακα για παράδειγμα. Ή βιοπανομοιότυπα. Δεν είναι εύκολη η ερευνητική μέθοδος. Εξασφαλίζει και ε, εποπτεία των βιοτεχνολογικών καταχωρήσεων αυτό μπορούν να το κάνουν και οι εθνικές υπηρεσίες και για τη συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς κυρίως με την, τον Αμερικανικό Οργανισμό FDA γιατί βρίσκεται στο, στο στόχαστρο για πολλά σκάνδαλα οπότε με βάση το TTIP και τις διαπραγματεύσεις που έχουμε για τη συνεργασία και τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτή τη στιγμή τι σχέση έχει η ΕΜΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με την FDA. Επίσης, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ε, τον κανονισμό και την οδηγία για τα ιατρικά, φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Και μάλιστα ε, ακούσαμε ότι για τα, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ασχολείται ε, η, η αίμα, αλλά θα είναι 5 έως 6.000 ε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα είναι πολύ λιγότερα. Είναι έτοιμη να αναλάβει τέτοιο έργο και τέτοιες προκλήσεις ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους όλων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, Αρχών και Κέντρων. Είναι πολύ καλό να έχουμε απευθείας ενημέρωση από εσάς. Όχι μόνο για να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η δουλειά σας, αλλά επειδή απευθύνατε και έκκληση ε, για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ως προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Νομίζω η αυξανόμενη σημασία αυτού του κέντρου αναδεικνύεται και με, στα πλαίσια αυτής της απειλής, που, της πίεσης που δεχόμαστε από τον έμπολα και την εξαπλωσή του. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ασχοληθούν και με την αναχέτηση της εξάπλωσης νόσου στην Ευρώπη, αλλά θα έπρεπε να εντείνουν και τις προσπάθειες τους ή τις δράσεις τους στο επίκεντρο εκεί που υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα της ασθένειας γεωγραφικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον ιό έμπολα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς απειλές θα έπρεπε να είναι αντικείμενο του οργανισμού σας, του κέντρου σας, αλλά για την ώρα χρειάζεται δική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στις 15 Οκτωβρίου Ακόμα συζητούσαμε πώ θα βοηθήσουμε στην αναχέτηση τη εξάπλωση του ιού στη Δυτική Αφρική. Γιατί, γιατί να μην υπάρχει απόσπαση ειδικών από τον ECDC ε για τρίτε χώρε εφόσον είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ή τέλο πάντων με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο να βοηθήσει έξω χώρε, χώρες, όπως η Μολδαβία ή και Ουκρανία, σε περιπτώσει που χρειάζονται αρρωγή και σε σχέση με όσα συμβαίνουν με τον νέο έμπολα και ένα χρόνο περίπου και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ήθελα να μου πείτε ο συντονίστρια το εξή. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή του χρόνου να οργανώσουμε μια κοινή συνάντηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και OCDC για να έχουμε μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων ε, και των επιπτώσεων τη σημερινή κρίση, αλλά και το τι μαθήματα αντλήσαμε από αυτή την κρίση και αν είναι πολύ σαφείς οι αρμοδιότητές σας θα είναι πολύ πιο σαφής η δράση που πρέπει να αναλάβουμε. Διότι αυτό που βλέπουμε από την τωρινή κρίση είναι ότι ενώ το κέντρο λειτουργεί μια χαρά, θα μπορούσε το πεδίο του να επεκταθεί και να απευθυνθεί και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεριξιστικά χρειάζονται βοήθειά του. Ευχαριστούμε ο κύριος Βελτιθίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των οργανισμών που ήρθαν εδώ και για τι παρουσιάσει τους. Είναι μεγάλη μα χαρά να υποφεληθούν τις ειδικέ τους γνώσει και μελλοντικά. Δύο ερωτήσεις για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Πρώτον, η διαδικασία διοδότησης για την έγκριση, μάλλον για την αποτελεσματικότητα ενό φαρμάκου ε, προβλέπει τα ίδια στάδια δοκιμής που προβλέπουν και μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Δηλαδή για τις περιπτώσεις που είναι κατεπίγουσες υπετρέπονται ειδικές δοκιμές, δοκιμές όπως ε, ε, για το φάρμακο που θα θέλαμε να αντιμετωπίσει τον ιό έμπολα. Επίσης για πολλά βιολογικά φάρμακα που έχουν ανακοινωθεί σε επαναστατική ανακάλυψη στον τομέα της ογκολογίας. Αυτά γίνονται αντικείμενο εμπορίας ή χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν αποδείξει την πραγματική του δραστικότητα. Όχι σε όλε τι περιπτώσει, κάπου την έχουν αποδείξει, αλλά συνήθω δεν έχουν δείξει να είναι πραγματικά δραστικά. Και πολλούνται πανάκριβα, ε, ενώ χρησιμοποιούνται ήδη στα νοσοκομεία. Υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσετε τη διαδικασία evidence-based medicine, φάρμακο βασιζόμενες αποδεικτικά στοιχεία. Ευχαριστούμε κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις προς τον Διευθυντή Ράζη. Πρώτα απ' όλα για την εσωτερική αγορά στην Ευρώπη και για τα φάρμακα. Εγώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχομαι από μια περιοχή παραμεθόριο, πολύ τουριστική. Υπάρχει ένα φαρμακείο και αν έρθει κάποιος τουρίστας από οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήσει ένα φάρμακο που έχει συνηθίσει να βρίσκει στη χώρα του, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να το, το πωλήσει γιατί απαγορεύεται. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρότατη φραγμή για την εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι γι' αυτό. Είναι απλώς ένας περιορισμός της εσωτερικής αγοράς για λόγους οικονομικούς. Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη, υπενηχθήκατε ότι υπάρχει θέμα με το κόστος των φαρμάκων. Και ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα. Όλο ένα και περισσότερο Εγκρίνεται και αδειοδοτείται φάρμακα στο Λονδίνο, δηλαδή έχουν ευρωπαϊκή άρια κυκλοφορία, που δεν μπορούν μετά να χορηγηθούν στους ασθενείς των κρατών μελών διότι είναι πολύ ακριβά. Οι εθνικές υπηρεσίες υγείας δεν δέχονται τη διανομή των φαρμάκων αυτών από τις υπηρεσίες τους διότι το κόστος δεν μπορούν να το καλύψουν. Εσείς τι ρόλο παίζετε από, για αυτές τις περιπτώσεις ε, από το Λονδίνο πώς ε, επηρεάζεται και έρχεστε στην επαφή με τις Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας. Ευχαριστούμε κυρία Καμπεθόν Ρουίς. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς την Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και χαίρομαι που εξακολουθεί να εμπίπτει στο θέμα της πρόσθεσης των καταναλωτών και όχι στη βιομηχανία, στην Επιτροπή Ένδη και όχι στην Επιτροπή Ήτρε. Είναι πολύ σημαντικές οι προκλήσεις του οργανισμού αυτού του ΕΟΦ, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για την ισότητα πρόσβαση στα φάρμακα και τη φαρμακευτική περίθαλψη, κυρίως πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα. Χαίρομαι που είναι από τις προτεραιότητες του οργανισμού η διευκόλυνση της πρόσβασης στα φάρμακα. Εξού και η ερώτησή μου. Τι γνώμη έχετε για το τι μπορεί να γίνει για να σταματήσουν κάποια μονοπόλια για συγκεκριμένα φάρμακα που έχουν αποφασιστική σημασία γιατί αφορούν πολύ σημαντικές ασθένειες. Και πώς θα σταματήσουμε την αδιαφάνεια στην διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών για τις καινοτόμες κυρίως θεραπείες. Επίσης, πώς θα εξορροπηθεί τεράστια διαφορά των τιμών φαρμάκων μεταξύ των διαφόρων χωρών πέραν της χρηματοδότησης της εθνικής για τα φάρμακα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση των τιμών φαρμάκων στις χώρες μέλη. Και αυτό φυσικά δυσχεραίνει την, το έργο της ΕΜΑ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, ένα φάρμακο για τη σκολικοειδίτιδα έχει πολύ σημαντική διαφορά στις τιμές. Πώς θα διευκολύνεται, παραλαμβάνω, την καλύτερη πρόσβαση στην καινοτομία, ιδιαίτερα για τις σπάνιες νόσους, που θα πρέπει να αποτελεί, και όπως είδαμε αποτελεί προτεραιότητα και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων. Επίσης, πώς θα καταπολεμήσουμε την ε, πώληση νοθευμένων ε, φαρμάκων που ε, έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα και κέρδη από ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών από έχουμε μάθει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στάς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση για την ΕΦΣΑ έχουμε να κάνουμε κι εμείς. Ε, διάφορες φορές ακούσαμε την ερώτηση αυτή για την ανεξαρτησία και τη σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγωνιστήκαμε και με τον προκάτοχό σα τα τελευταία χρόνια. Πολλά διάφορα έγιναν Προ το καλό. Το αναγνωρίζουμε. Εξακολουθεί να υφίσταται όμως η ανησυχία όχι μόνο από ΜΚΟ και η διαμεσολαβήτρια ε, πρόβαλε διάφορα στοιχεία. Ο τύπος επίσης ε, έκανε αναφορά για διάφορα πράγματα που πήγαν στραβά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια σειρά γεγονότων περιστατικών που υποδεικνύουν ότι διάφοροι επιστήμονες έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τη βιομηχανία και ότι ουσιαστικά ακολουθούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Πώς θα συνεχίσετε λοιπόν τις προσπάθειες οι οποίες ε, ομολογουμένως κινούνται, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά μια μη κυβερνητική οργάνωση που δημοσίευσε μια μελέτη για την ε, χειραγώγηση στοιχείων σε ό,τι αφορά το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Γνωρίζετε τις ε, αιτιάσεις που εκφράστηκαν. Θα τις εξετάσετε, θα απαντήσετε. Θα με ενδιαφέρει κύριε να ακούσω την απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του ομιλητέ. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση. Γιατί ξεκινήσαμε τόσο καθυστερημένα για το εμβόλιο, με το εμβόλιο για το έμπολα. Πολύ σημαντική ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Σπρίνγκερ. Θεωρώ ότι η οργάνωσή σας κάνει πολύ καλό έργο. Το ήξερα. Μάλλον με το ήξερα στο παρελθόν, το παρακολουθώ από τον Ιούνιο όμως ο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καλός. Και τι γίνεται με την Αφρική, σημαντικό. Και τρίτη ερώτηση. Κάθε χώρα θέλει να πετύχει καλά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε. Και τρέλο, σε ό,τι αφορά την ΕΦΣΑ, πολύ σημαντικά αυτά που κάνετε, αλλά ποιον καθοδηγείτε τελικά. Τέλος, λέει ο Πρόεδρο, ο κ. Κρότε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει για τον κ. Ράση. Καταρχά, Και όντω ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν επικαλύψεις. Ποια είναι ο συντονισμό μεταξύ των οργανισμών, ποια μέσα υπάρχουν για να γίνονται συμφωνίες στον κύριο Ούλου. Η Πάρμα δεν είναι και ομφαλός του κόσμου. Συζητείτε ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Τι κάνει ένας επιστήμονας που πηγαίνει στην Πάρμα για τρεις ημέρες όταν φεύγει για τρει ημέρε δηλαδή από τη βιομηχανία στην οποία εργάζεται. Πώ ζητάμε δηλαδή από του εμπειρογνώμονε καταρχά να είναι εκεί, να είναι στην ε, εχμή του δόρατο, αλλά παρόλα αυτά να είναι και ανεξάρτητοι. Πώ το πετυχαίνετε αυτό το αδύνατο γιατί συχνά κατηγορείται η ΕΦΣΑ και όλοι οι οργανισμοί ότι παίρνει τους πιο καλούς εμπειρογνώμονες, τους πληρώνει για ένα μηταμινό ποσό για τρεις ημέρες ε, που τους βγάζει από την κανονική τους δουλειά. Πώς ε, καταφέρνουμε λοιπόν να τραγωνίσουμε τον κύκλο, για εξηγήστε μας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Να ζητήσω από όλους τους εκτελεστικούς διευθυντές να είναι πάρα πολύ σύντομοι, γιατί θα πρέπει σε 10 λεπτά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις απαντήσεις και τις τρεις απαντήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη και στις 6.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει με μία μικρή ευελιξία. Και μετά θα... Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ίδια σειρά. Να δώσουμε το λόγο στην ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλέ ερωτήσει και πολύ ενδιαφέρον για το έργο τη ΕΦΣΑ, Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων. Κυρία Γιούζο, ναι, θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία με του ετούντε και ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουμε ακριβώ αυτή την επικοινωνία, το διάλογο με τους ετούντες, χωρίς φυσικά να διακυβεύουμε ή να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία και την ποιότητα του ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων. Για τη συνεργασία. Συνεργασία οργανισμού και επιστημόνων. Έχουμε 470 ανθρώπους προσωπικό, οι μισοί είναι επιστήμονες το μισό προσωπικό του οργανισμού. Έχουμε και πάνελ και ομάδες εργασίας, 10 πάνελ από 21 επιστήμονες και επιπλέον 200 μέλη πάνελ 1500 ε, εμπειρογνώμονες ε, έχουμε που συνεργάζονται μαζί μας σε διάφορες ομάδες εργασίας. Και επίση ζητούμε συγκεκριμένα δεδομένα. Απευθύνουμε κλήσει για συλλογή δεδομένων και η κοινωνία των πολιτών, οι ακαδημαϊκοί κύκλοι, πανεπιστημιακοί, εταιρείε μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την έκκληση που απευθύνουμε. Τώρα, για τους χειρισμούς υγείας. Έχουμε εκδώσει πάνω από 570 επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στην ιστοσελίδα μας και μόνο για τους οργανισμούς υγείας. Θα τους βρείτε στον ιστότοπό μας. Επίσης, αν έχουμε αρκετούς ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες, επιστήμονες. Φυσικά και έχουμε, ε, γιατί κάθε τρία χρόνια έχουμε ένα ανοιχτό διαγωνισμό. Περίπου χίλιες αιτήσεις λαμβάνομαι από επιστήμονες. Και κάνουμε μια αξιολόγηση ανάλογα με, την, ε, με τα προσόντα τους. Φυσικά εξετάζουμε τα ενδιαφέροντά τους και κατά πόσο διαπιστώνουμε μία σύγκρουση συμφερόντων ε, και αποκλείουμε τους επιστήμονες για τους οποίους ε, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και σας διαβεβαιώ και το λέω και στον κύριο Γκρότε, πώς θα έχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη και ταυτόχρονα ανεξαρτησία. Όντως είναι δύσκολο, είναι πρόκληση, αλλά ακριβώ με τον ανοιχτό διαγωνισμό που κάνουμε κάθε τρία χρόνια και με το στιβαρό σύστημα αξιολόγηση ε, και διαχείρισης ε, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων έχουμε αποδείξει τα τελευταία, τελευταία χρόνια ότι το σύστημά μας είναι αποτελεσματικό. Τώρα, αν είναι τέλειο, όχι τέλειο δεν είναι, μπορεί να βελτιωθεί. Θα το βελτιώσουμε μάλιστα, θα προσθέσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερο άνοιγμα για να συμπληρώσουμε την πολιτική μας σύγκρουση συμφερόντων με μεγαλύτερη διαφάνεια και άνοιγμα. Αλλά φυσικά για μερικά μέλη των πάνελ ίσως είναι ρευστά τα όρια. Άλλωστε δεν αποφασίζει μόνο ένας επιστήμονας, ένας εμπειρογνώμονας ένα πάνελ, αλλά 21. Οπότε ακόμη και αν υπάρχει σύγκρουση για τον έναν, δεν θα επηρεάσει την απόφαση γιατί είναι συλλογική. Έχουμε το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα και για την καινοτομία και έχουμε τις δοκιμές που κάναμε και για το πρόγραμμα Grace θα βρείτε τα αποτελέσματα στο, στην ιστοσελίδα. Κύριε Στάσαν, έχουμε εχέγγυα. Νομίζω ότι το σύστημα μας έχει εχέγγυα για τη σωστή αξιολόγηση, για τη σύγκρουση συμφερόντων και επαναλαμβάνω το σύστημα το βελτιώνουμε διαρκώς. Δεν συμφωνώ ότι οι επιστήμονές μας προέρχονται από τη βιομηχανία. Εμείς επιλέγουμε τους επιστήμονες με βάση την ανεξαρτησία τους και φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε την αμεροληψία τους. Τώρα, αν έχουμε νέα επιστημονικά απορίσματα για το ΜΟΝ 810, για παράδειγμα, τη νέα ποικιλία γενετικώς τροποποιημένου καλαμποκιού, τότε ξανανοίγουμε τη διαδικασία για τη μελέτη επιπτώσεων. Συνεχώς λαμβάνουμε υπόψη τα νέα επιστημονικά πορίσματα και τις νέες επιστημονικές γνώσεις. Ευχαριστώ. Κύριο Σπρέγκερ από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα, το, ε, την υπεύθυνη για την επαφή με την ομάδα ΕΜΒΗ. Ναι, προσφέρουμε στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή έχει επιτρέψει την αποστολή ειδικών προς τη Δυτική Αφρική. Έχουμε όμως πολλά αιτήματα για πρόσθετη στήριξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς είναι καλό στο μέλλον να κοιτάξουμε να συζητήσουμε αν υπάρχει ανάγκη ή επιθυμία ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσεων να παράσχει περισσότερη στηρίξη σε χώρε εκτό ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Νομίζω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία που μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά αυτό θα απαιτήσει και πρόσθετου πόρου. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση τη κυρία Φένερ Πίρικ, νομίζω ότι Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ καλή η διαδικτύωσή μα με την Επιτροπή Ασφάλεια και Υγεία Τώρα, για την ερώτηση, ε, τη συγκεκριμένη που μου κάνατε, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είναι εκτό του του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Ευχαριστούμε και τώρα τελευταίος ο κύριος Ράζη. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γιατί έχω κάμποσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις ε, ομαδοποιήσω αντί να τις απαντήσω μία-μία. Η πρώτη έχει να κάνει με τις βιοτεχνολογίες. Εάν τις αποτιμούμε εμείς οι ίδιοι, περιμένουμε και την ε, εθνική έγκριση. Οι βιοτεχνολογίες ε, και τα βιοφάρμακα ε, ελέγχονται και εγκρίνονται μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Βεβαίω, αν είναι συσκευέ για το βιοτεχνολογίε, είναι πολύ περίεργο όρο. τότε τις τι εγκρίνουν οι εθνικέ υπηρεσίε. Για τον αίμα και τη συνεργασία του με τον EFMA έχουμε μόνο τεχνική συνεργασία, δεν υπάρχει διμερής ε, συμφωνία. Υπάρχει μάλιστα μια σχέση απορρίτου, κυρίως για σκοπούς εμπιστευτικότητας, ποιότητας. Έχουμε κάποια πολύ καλά παραδείγματα που μας ενημέρωσαν Και όλο το δίκτυο φαρμακοπαγρύπνηση στην Ευρώπη αμέσως κινητοποιήθηκε για να είμαστε σε επιφυλακή. Επίσης με το νεό έμπολα είχαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις και προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε κάπως τις διαδικασίες ώστε να μην προκαλέσουμε σύγχυση στο κοινό για κάτι που εγκρίνεται από εμάς και όχι στις ΗΠΑ και αντιστρόφως. Ε, για να αισθάνονται άνετα οι ασθενείς ως προς το τι γίνεται στις περιοχές της παραμεθόριας, κοντά στα σύνορα και τι γίνεται για κάποιον που δεν μπορεί να πάρει ένα φάρμακο για λίγα χιλιόμετρα απόσταση στην Ευρώπη. Ναι, ε, τέτοια αποδεκτικά στοιχεία δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Διότι η εθνική νομοθεσία πριτανεύει. Εμείς μπορούμε να δώσουμε σε ένα φαρμακό τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Αφού δώσουμε αυτή την άδεια όμως, κάθε κατός μέλος μπορεί να διαθέσει το φάρμακο αυτό. Αλλά το πώς θα γίνεται η επιστροφή. Ε, του κόστους ή πώς θα συνταγογραφείτε, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών Δεν μπορούμε να παρέμβουμε καθόλου. Ε, <clears throat> και αυτό με φέρνει στο ευρύτερο θέμα της τιμής και της διαθεσιμότητας. Η πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε την ερχόμενη πενταετία είναι ακριβώς αυτή νομίζω. Διότι μετά από 20 χρόνια ε, επιτυχημένης κεντρικής αδειοδότησης και έγκρισης, το θέμα είναι τώρα εάν πια οι, οι τιμές αυτές ε, είναι προσιτές. Οι τιμέ δεν είναι ένα τομέα που μπορούμε να επηρεάσουμε, δεν έχουμε καμία σχετική αρμοδιότητα. Όμω κάποια πρωτοβουλία για να επηρεάσουμε αλλιώ ίσω να μπορούσε να γίνεται. Είπα και στην παρουσίασή μου ότι απευθυνόμαστε στου φορεί που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση τεχνολογιών τη υγεία και του ε, ε, φορεί που καλύπτουν τα έξοδα στα κρατημέλη. Αυτό σημαίνει ότι για την σχέση κόστους ωφελίας για την αποτελεσματικότητα και την δραστικότητα των φαρμάκων μπορούμε να ενημερώνουμε και αυτό θα μπορούσε να γίνεται εκ παραλίλου και όχι διαδοχικά δηλαδή να, εκτιμά, να συναποτιμάται για την, η δραστικότητα του φαρμάκου μαζί με τη δυνατότητα των ε, αρχών που επιστρέφουν ε, το κόστος ε, να καλύψουν το κόστος αυτό. για την ώρα, λόγω της καλής μας διάθεσης και λόγω καλής, βάσει της καλής μας πίστης μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά μαζί τους. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές για να ε, με την προσαρμοστική αδειοδότηση adaptive licensing το έχουμε ονομάσει ε, ελπίζουμε αν αυτό εφαρμοστεί πλήρως να βελτιώσει τα πράγματα και ένα επιπλέον λεπτάκι παρακαλώ. Για τον ιό έμπολα. Για το εμβόλιο να πω ότι δεν έχουμε καθυστερήσει. Τα εμβόλια και το ακούω από τους παραγωγούς λένε ότι δεν ότι έχουν κάτι στα σκαριά, αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα έτοιμο. Υπάρχει ταχεία διαδικασία και θα ενεργοποιηθεί εάν έχουμε το παραμικρό δεδομένο. Όπως προείπα, έχουμε με τουλάχιστον τρεις ε, παραγωγούς εταιρείες επαφές δεν θα τους βάλουμε να περιμένουμε, θα υπάρχει ταχεία διαδικασία, αλλά χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Μόλις έχουμε τα δεδομένα στη διάθεσή μας θα σας πούμε περισσότερα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω όλους. Με συγχωρείτε, ξέχασα μία. Ναι, ναι, πώς συνεργαζόμαστε. Ε, δεν ε, ε, ε, ξέρω αν εννοείται μεταξύ μας ή με τις εθνικές αρχές. Μεταξύ μας είναι πολύ απλό. Διεπόμεθα από την ίδια νομοθεσία και λειτουργούμε βάσει της ίδιας διαδικασίας. Ως τώρα δεν είχαμε κανένα σοβαρό πρόβλημα, αντιθέτως είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε τα επιστημονικά μας στοιχεία, ιδίω ε, βάσει των νομοθετικών εργαλείων. Μεγαλύτερη δυσκολία υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Με προϊόντα που δεν ε, καλύπτονται σε κεντρικό επίπεδο αυτό. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα αμέσως, αμέσως πρέπει να περάσουμε στο σημείο 7. Απευθείας θα περάσω στον εκπρόσωπο τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Μάικλ Σκάνελ από το Γραφείο Τροφίμων και Εκτενιατρικών Θεμάτων. Και μετά θα δούμε την ερώτηση των συναδέλφων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί έχει περάσει και η ώρα. Το Γραφείο Τροφίμων Εκτενιατρικών Θεμάτων ιδρύθηκε το 1997. Και το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ίδρυσής μας είναι ότι ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έγινε λοιπόν μελέτη και έρευνα του Κοινοβουλίου και μία από τις βασικότερες Ένα λοιπόν θέμα της ε, σπογγόλου εγκεφαλοπάθειας ήταν ότι έλειπε ένας μηχανισμός ε, ο οποίος θα διασφάλιζε ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους με υψηλό επίπεδο εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πόρισμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε αποδεκτό από το, το, την Κομισιόν και θυμάμαι τον Πρόεδρο Πρώτη και την επιβεβαίωση του Σεπτέμβριου του 1999 εδώ στο Κοινοβούλιο που έθεσε το πολύ καλό ερώτημα του γιατί η Ευρωπαϊκή ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έπρεπε να εμπιστευτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω διευρύνσει, αν δεν μπορούμε να πετύχουμε την ασφάλεια τροφίμων. Είναι κάτι τόσο βασικό. Έγινε λοιπόν πολύ έλεγχη σε πολλές χώρες και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί το μόντζο πράντι μας. Κάνουμε επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που εφαρμόζεται, που ισχύει, εφαρμόζεται σωστά πώς το πετυχαίνουμε και τι θέματα ερευνάμε. Καταρχάς, κοιτάμε την ίδια την νομοθεσία. Προφανώς, αν δεν έχει μεταφερθεί, δεν έχει νόημα να κοιτάξουμε τα υπόλοιπα. Ελέγχουμε αν υπάρχει αρμόδια αρχή, αν υπάρχει καλός συντονισμός σε όλο το φάσμα ελέγχων και ότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος και η ευθύνη τους ελέγχουμε κατά πόσον υπάρχει επαρκές προσωπικό για να κάνει τους ελέγχους, αν υπάρχουν επαρκή άτομα, αν έχουν τα σωστά προσόντα, τη σωστή εκπαίδευση, αν η αρμοδία αρχή έχει τις εξουσίες να διεξαγάγει τις, ε, τα καθήκοντά της, το ρόλο της, ε, αν έχει για παράδειγμα άδεια εισόδου στις επιχειρήσεις τροφίμων, αν έχουν αρμοδιότητες να επιβάλλουν περιορισμούς, να κλείσουν επιχειρήσεις. Κοιτάμε επίσης κατά πόσον γίνονται έλεγχοι επιθεωρήσεις αξιοποιώντας σωστά τους πόρους και κατά πόσον επικεντρώνονται στα σωστά σημεία, κατά πόσον έχουν αρμοδιότητες να επιβάλλουν κυρώσεις, οι οποίες να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, το οποίο στην πράξη μπορεί να αποβεί δύσκολο. Ελέγχουμε κατά πόσον υπάρχει απαραίτητη υποδομή για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αυτό περιέχει για παράδειγμα τα εργαστήρια. Και σε ό,τι αφορά τις κάτω πήγουσες ε, ε, περιπτώσεις ε, και τις επιζώτιες, κοιτάμε κατά πόσο υπάρχει σχέδιο κατά πήγουσες ανάγκης. Γιατί αν δεν είναι προετοιμασμένος κανείς για κρίση, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με σωστό τρόπο. Και επειδή κάθε κρίση έχει διαφορετικό πρόσωπο, πρέπει να υπάρχει πολλή προετοιμασία προκειμένου να μπορεί κανείς να αντιδράσει αποτελεσματικά. Ένας άλλος βασικός στόχος του ρόλου μας είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί αν σε μια κοινότητα των 28 κρατών μελών υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο αποτελεσματικότητας, μάλλον σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι οι διαφορές αυτές ε, υπονομεύουν το συνολικό επίπεδο ελέγχου και αποτελεσματικότητας και οι φορείς και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη ότι υπάρχει σωστό επίπεδο ελέγχου σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ βασικό για την ενιαία αγορά και τη λειτουργία της και αποτελεί και το μέτρο της απαντητικότητας όλων των μέτρων μας. Μπορούν οι επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη και οι τρίτες χώρες να είναι σίγουρες ότι υπάρχουν έλεγχοι σε αποδοτικό επίπεδο, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει ενιαία αγορά και σε έναν τομέα τόσο σημαντικό πολιτικά αλλά και οικονομικά όπως το τρόφιμα, αυτό έχει σοβαρότατες συνέπειες. Και ύστερα γενικά τα αποτελέσματα είναι θετικά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Και αυτό με τη σειρά του αποτυπώνεται με την έλλειψη μονομερών μέτρων ε, ασφαλιστικής δικλίδας. Υπήρχε μια εποχή στην ε, Ευρώπη όπου τα κρατημέλη επέβαλαν με το παραμικρό μονομερείς ε, κυρώσεις, μονομερείς πληρισμούς. Και αυτό συχνά γινόταν για προστατευτικούς σκοπούς, σκοπούς προστατευτισμού. Αυτό τώρα έχει εκλείψει ως επιτοπλίστων. Παρουσιάζονται που και που προβλήματα, αλλά γενικά τα κρατημέλη εμπιστεύονται και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη χωρίς να λαμβάνουν μονομερή μέτρα. Έχουμε λοιπόν σωστά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Επειδή δεν έχουμε και χρόνο, Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ε, δύο λόγια. Εμείς ε, δεν είμαστε οργανισμός, είμαστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά σήμερα εργαζόμαστε σε νέους τομείς, σε ό,τι αφορά τις ιατρικές συσκευές, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το σκάνδαλο. Το πρόσφατο, ε, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρχές ιατρικών συσκευών στα κρατη και κάναμε διάφορες επιθεωρήσεις σε όλη την Ευρώπη για να υπάρχει εμπιστοσύνη στον τομέα των ιατρικών συσκευών σε ό,τι αφορά γεωγραφικέ γεωγραφικές ενδείξεις, ε, τα σήματα, τα συστήματα τα οργανικά, τα βιολογικά. Και τέλο, για να κλείσω, επειδή ε, ενώ δεν είμαστε οργανισμό ξεχωριστό, παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το Κοινοβούλιο. Γιατί, όπω σα είπα και προηγουμένω, ε, το Κοινοβούλιο ουσιαστικά μα ίδρυσε και είμαστε διτεθειμένοι να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερω με τον συντονιστή κύριο Στάσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Στάις που είναι ο άνθρωπός μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η λειτουργία του οργανισμού του γραφείου είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Όλες οι μελέτες και οι εκθέσεις επιθεωρήσεων διατίθενται στο διαδίκτυο. Το μόνο που λείπει θεωρώ από δικής μας πλευράς είναι η πολιτική παρακολούθηση των ε, θεμάτων. Συχνά παρακολουθούμε τα θέματα αυτά μόνο όταν ξεσπάει κάποιο σκάνδαλο. Εγώ θα ήθελα μαζί με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να παρακολουθούμε τι λειτουργίες και τον αντίκτυπο των συστάσεων του Γραφείου Τροφίμων και Εκτινωτικών Θεμάτων προκειμένου να υπάρχει και πολιτική συνέπεια. Και κάτι άλλο. Είναι εποχή α, ε, περικοπών. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό αλλά γνωρίζοντας το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινωτικών Θεμάτων, μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι τα 190 άτομα τα οποία δουλεύουν στο γραφείο αυτό πραγματικά χρειάζονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία εκεί. Με πιο λίγα άτομα θα είναι πολύ δύσκολο η διεξαγωγή του έργου του Και εδώ πέρα θα κλείσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Σέκπερικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη Πρόεδρε γιατί η οργάνωσή σας ε, τη γνωρίζω και από το Κοινοβούλιο της ε, Ολλανδίας. Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε θέματα αντιβιωτικών βλέποντας τι γίνεται η Ολλανδία είναι πάρα πολύ αυστηρή, άλλες ε, χώρες δεν το κάνουν αυτά και τελικά είμαστε τα θύματα. Σε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις βαλβίδες για τους χείρους. Η Ολλανδία τα κάνει όλα αυτά, κάποιες άλλες χώρες όχι. Κάποιες χώρες λοιπόν ε, εφαρμόζουν αυστηρά κάποια ζητήματα, ενώ κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο χαλαρές. Και αυτό ισχύει και κατεξοχήν για τα αντιβιωτικά. Δεν έχω άλλον κανέναν που να ζητάει το λόγο, οπότε να επιστρέψω στον, ε, στο γραφείο των ε, κοινωνικών θεμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, δύο μιλητές. Κύριε Στάς, πολύ ευχαρίστως να αποδεχτώ την πρόσκληση να έχουμε ετησίως μια συνάντηση για να παρουσιάζουμε το έργο μας και να απαντούμε σε απορίες και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Για το θέμα των πόρων δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε τους πόρους μας, αλλά γίνονται πολλές οικονομίες. Γιατί δεν θα κάνουμε όπως μερικοί άλλοι που ακόμη και σε περίοδο ε, ένδυας δημοσιονομικής ε, διεκδικού νέου πόρου. Δεν κρυβόμαστε πίσω από ε, το, επιχείρημα της έλλειψης πόρων. Ε, εδώ χρησιμοποιούμε ως άλοθη για να μην ανταποκρινόμαστε στο έργο μας. Το κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους πόρους μας. Τώρα, θέλουμε να διασφαλίσουμε φυσικά παρά τις διαφορές στο επίπεδο εφαρμογή που υπάρχει, δεν θέλουμε μια κατάσταση που να υπονομεύει την υγεία ή την αξιοπιστία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την, ε, ακόμη και στην περίπτωση διαφορών και διαφορετικών επιδόσεων, θέλουμε ακόμη και οι κακοί μαθητές, οι χειρότεροι μαθητές, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Γι' αυτό έχουμε στοχευμένες συστάσεις, έτσι παρακολουθούμε με πολύ διαφανή τρόπο. Έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε χώρα και γνωρίζουμε που υπάρχουν αδυναμίε και που δεν σημειώθηκε ιδέω πρόοδος. Και μια νέα κάτι καινοτόμο είναι η εκθέσεις επισκόπησης, γενικής επισκόπησης, όπου εξετάζουμε την κατάσταση σε συγκεκριμένου κράτου σε όλα τα κράτη-μέλη, εντοπίζοντα τι αδυναμίε, τι ελλείψει και προτείνοντα τρόπου για την διόρθωση. Για το θέμα των αντιβιωτικών, ε, το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά, ε, το περιλάβαμε ιδιαίτερα στις αποστρέψεις που είχαμε για το κρέας πουλερικών. Ε, είχαμε Συγκεκριμένε προτάσεις προ τα κράτη-μέλη για να ε, μειωθεί αυτή η αντοχή στα αντιβιωτικά. Και επίση είχαμε μια ε, διυπηρεσιακή ομάδα για το θέμα της μικροβιακής αντίστασης, ε, της αντίστασης στα αντιβιωτικά και προσπαθούμε και αυτό το σημείο να το συμπεριλάβουμε στον τακτικό μας έλεγχο. Σας ευχαριστούμε θερμά και να ευχαριστήσω και τον εκτελεστικό διευθυντή, τους εκτελεστικούς των διαφόρων οργανισμών και τον ε, πρόεδρο του γραφείου για τα κτηνιατρικά θέματα και τα τρόφιμα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνεδρίαση και να σας προσκαλέσω σε μια δεξίωση. Θα λάβει χώρα ακριβώς έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.